Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να απολογηθώ για την καθυστέρηση, αλλά υπήρξε μια μικρή, θα έλεγα, σύγχυση ε, με το Προεδρείο και πρέπει να σας πω ότι τώρα έχω ειδοποιηθεί για να είμαι εδώ. Όμως θα προχωρήσουμε τη διαδικασία όσο γίνεται πιο σύντομα και με γρήγορους ρυθμούς. Για άλλη μια φορά απολογούμε εκ μέρους της Επιτροπής. Mr. Tavares, Rapporteur of the Review of the EU's Human Rights Strategy κύριος Ταβάρες ο εισηγητής για την ανθεώρηση στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου συμφώνησε η έκθεσή του να συζητηθεί πριν από την ενημέρωση από την κυρία Ερατό Κοζάκο Μαρκουλή, την Υπουργό Εξωτερικών, η οποία μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της 15ης ε, Οκτωβρίου ταυτόχρονα η έκθεση της κυρίας Χάκε ε, αναβάλλεται. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Στο Πού I have the pleasure of Έχω την χαρά να παρουσιάσω την κυρία Σάρα Κλίφ αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΙΕ σχετικά με την υποστήριξη χωρών που βρίσκονται υπό μεταβατική φάση. Με στόχο την πρωτοβουλία του ΙΕ για την ανάπτυξη συνεργασία μετά τι συγκρούσει. Η κυρία Κλήφη ασχολείται με πέντε τομεί. Τι πολιτικέ διαδικασίε, την ασφάλεια, δικαιοσύνη, οικονομία, νομοθεσία και λειτουργικότητα της διοίκησης. Ξανά απολογούμε γιατί χάσαμε ένα αρκετό χρόνο. Κυρία Κρύφ. Thank you very much, Chair. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε μέλη της Επιτροπής για την ευκαιρία που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα των μη στρατιωτικών ικανοτήτων. Στρατιωτικές ικανότητες είναι μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ που ξεκίνησε από κάτι σημαντικό που συνειδητοποιήσαμε, ότι δηλαδή εάν δεν μπορούμε να στηρίξουμε σημαντικά και ισχυρά στιβαρά θεσμικά εθνικά όργανα, κάτι το οποίο όπως είπε και ο Πρόεδρο δίνει στον κόσμο την έννοια τη πολιτική εκπροσώψης, αλλά και αστυνομία που του προστατεύει, δικαιοσύνη και δικαστέ που του δίνει το αίσθημα τη δικαιοσύνη, οικονομικά θεσμικά όργανα τα οποία παρέχουν τα βασικά της οικονομίας και της εργασίας. Εάν δεν μπορούμε λοιπόν να στηρίξουμε αυτούς τους θεσμούς σε χώρες οι οποίες βγαίνουν από συγκρούσεις, τότε τα προγράμματα αυτά ανάκαμψης δεν θα επιτύχουν. Με άλλα λόγια, συνειδητοποιήσαμε πως η στήριξη στα εθνικά στου εθνικού θεσμού σε χώρες όπως η Λιβύα, η Εμένη, Ακτή του Λεφαντοστού, Λιβερία, Αϊτή, Ανατολικό Τιμόρ, είναι βασικό κομμάτι των προσπάθειών μας και σημαντικό συμπλήρωμα της πολιτικής διαμεσολάβησης και των προσπαθειών ειρήνευσης που παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο συγκρούσεις αλλά από μόνες αυτές τις προσπάθειες δεν αρκούν έτσι ώστε οι χώρες να μην ε, κινδυνεύουν από το να υποτροπιάσει μια σύγκρουση. Αυτό λοιπόν καλύπτει η πρωτοβουλία μας, όπως είπε και ο πρόεδρος στην εισαγωγή του καλύπτει πέντε τομείς εθνικών ικανοτήτων σε χώρες όπως αυτές που ανέφερα, δηλαδή πολιτικές διαδικασίες, ασφάλεια, κράτος δικαίου, οικονομική αναδιοργάνωση και βασική διοίκηση. Είναι επίσης μια πρωτοβουλία η οποία αντλεί διδάγματα τα οποία μάθαμε με οδυνηρό τρόπο στην διεθνή κοινότητα από επανειλημμένες ειρηνευτικές αποστολές στην Αϊτή και στο Τιμόρ, τις δυσκολίες που συναντήσαμε στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Κάποια από αυτά τα μαθήματα ήταν η δυσκολία του να φέρνουμε κάποια τεχνικά μοντέλα από έξω σε κάποιες κοινωνίες, μοντέλα τα οποία όσο καλά και αν ήταν δεν μπορούν να μεταφυτευθούν ε, και οι θεσμοί από τη μία χώρα στην άλλη. Η δυσκολία επίσης του να ανταποκρινόμαστε αρκετά γρήγορα όσον αφορά την οικοδόμηση μη στρατιωτικών ικανοτήτων έτσι ώστε οι χώρες αυτές που βρίσκονται σε μετάβαση να έχουν την εμπιστοσύνη των πολιτών τους. Και επίσης να υπάρχει και η απαραίτητη εμπιστοσύνη και υπομονή ε, στις χώρες ε, αυτές ε, γιατί βεβαίως εμείς απ' έξω έχουμε πιο γρήγορα χρονοδιαγράμματα και προσδοκίες. Οπότε η πρωτοβουλία αυτή κάνει ουσιαστικά τρία πράγματα. Εργαζόμαστε σε κάποιες χώρες για να στηρίξουμε τις συγκεκριμένες χώρες. Έχουμε σχέσεις συνεργασίας για την παροχή εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης και υποστηρίζουμε την μεταρρύθμιση εντός του συστήματος του ΟΗΕ. Θα αναφέρω λοιπόν αυτούς τους τρεις τομείς έτσι γρήγορα και να αναφέρω και κάποια ζητήματα που προέκυψαν στις συναντήσεις μας εδώ πέρα τα οποία αποτελούν κοινέ προκλήσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά λοιπόν την εμπλοκή στις χώρες, το τελευταίο έτος στηρίζουμε την μετάβαση στην Λίβια, στη Λιβερία, στην ακτή του Ελεφαντεστού, στο Νότιο Σουδάν, την Αϊτή και στο Ανατολικό Τιμόρ. Επίση ε, ξεκινάμε να στηρίζουμε και τη μετάβαση της Ιεμένης και η συνάδελφος που μαζί μου σήμερα ήταν ε, και στην Συρία υπό διάφορες ιδιότητες. Κάποια μαθήματα λοιπόν τα οποία προέκυψαν είναι σημαντικά και για τον ΟΗΕ και για εσάς ε, όσον αφορά το πώς σκεφτόμαστε την στήριξη δημιουργίας θεσμών. Το πρώτο ήταν η ανάγκη στο να συνδυάσουμε τα μέσα πολιτικής και ασφάλειας για να υπάρξει μια συνοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαν υπάρξει προσπάθειες επί σειρά ετών στη Λιβερία να στηρίξουμε τις αστυνομικές δυνάμεις και δικαστήρια τα οποία θα δημιουργούσαν μια εσωτερική ασφάλεια με τρόπο μόνιμο. Οι προσπάθειες όμως αυτές είχαν αποτύχει διαφορετικές φορές για διαφορετικούς λόγους γιατί υπήρχαν και ειρηνευτικέ προσπάθειες για να οικοδομηθεί μια αστυνομία, η οποία δεν είχε, προσπάθεια η οποία δεν είχε συνδυαστεί, παραδείγματος χάρη, με τις προσπάθειες οικοδόμησης της δικαιοσύνης. Γιατί και όταν έγιναν αυτά τελικά δεν υπήρχε μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός για να πληρωθούν οι μισθοί των αστυνομικών και των δικαστικών που θα έπρεπε να εργαστούν. Οπότε συνεργαστήκαμε και με την πλευρά της λεγόμενης ανάπτυξης και με την πλευρά της λεγόμενης ασφάλειας για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση της Λιβερίας να καταρτήσει μια στρατηγική η οποία θα συνδυάζει αυτές τις πτυχές. Αστυνομία, δικαιοσύνη, σοφρονισμός, αλλά να υπάρχει και προϋπολογισμός μακροπρόθεσμος μέσω συνεργασίας και με των προγραμμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ. Ένα από τα δεύτερα, το δεύτερο δίδαγμα είναι πως χρειάζεται να υπάρξει μια διάρθρωση χρονική του προγράμματος μας για να λάβουν υπόψη την πολιτική πραγματικότητα στις χώρες αυτές. Τα μέλη της Επιτροπής σας φαντάζομαι θα το ξέρουν πως η πολιτικοί κύκλοι λήψης αποφάσεων συχνά είναι πολύ μακροσκελής και πολύ περισσότερο σε χώρες που έχουν περάσει μια κρίση όπου η πολιτική ηγεσία δεν είναι έμπειρη στη διοίκηση και έχουν δικά τους ζητήματα εμπιστοσύνης καθώς έχουν μόλις βγει από σύγκρουση. Οπότε ε, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Παραδείγματος χάρη στην ε, Λιβύη έχουμε μία προσέγγιση σε φάσεις. Δηλαδή λέμε πως πρέπει να υπάρξουν κάποιες βασικές ικανότητες γρήγορα, αλλά αναγνωρίζουμε πως θα χρειαστεί λίγος χρόνος για τους Λίβιους να πάρουν να περάσουν σε μια δική τους διαδικασία λήψη αποφάσεων για να μπορούν να μας πούνε τι στήριξη θέλουν. Οπότε αυτή η φάση της βοήθειάς μας είναι μια δεύτερη φάση προγραμματισμού. Ε, το τρίτο κύριο μάθημα που είναι πάλι σημαντικό για τον ΟΗΑ αλλά ίσως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το ενδιαφέρον για συνεργασίες για να οικοδομηθούν ικανότητες που συμπεριλαμβάνουν και βόρειες και νότιες χώρες. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης και τη μετάβαση την οποία περνάνε. Σε αυτές τις χώρες υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την εσωτερική εμπειρία μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε όταν κοιτάνε, ε, παραδείγματο χάρη το τι κάνουν με την κληρονομιά κάποιων δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες δεν θεωρείται ότι εξυπηρετούσαν ολόκληρο τον πληθυσμό, αλλά ήταν μέσω ενός αυταρχικού καθεστώτος και κοιτάνε παραδείγματο χάρη τον ε, έλεγχο, το πώς θα έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Έχουν εκφράσει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον για την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και μεταβάσεις όπως ε, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ε, στο παρελθόν. Έχουν επίσης εκφράσει το πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να έχουν βοήθεια από τη δική τους περιοχή του κόσμου με αραβόφωνους γιατί βεβαίως οι άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι μιλάνε αγγλικά ή γαλλικά είναι λίγοι σε αυτές τις κοινωνίες και με γνώση του τοπικού πλαισίου. Οπότε <coughs> αυτό το οποίο κάνουμε ως προσέγγιση βλέπουμε τη σημασία του πώς θα έχουμε κάποια βοήθεια η οποία θα συνδυάζει χώρες από τον Βορρά και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μεγάλη εμπειρία στην οικοδόμηση θεσμών ε, και υγιούς ε, διακυβέρνησης αλλά να τις συνδυάσουμε και με τις γειτονικές χώρες των χωρών αυτών που είναι υπομετάβαση και γνωρίζουν το τοπικό πλαίσιο και την πραγματικότητα κατόπιν οποίο εμείς που είμαστε πιο μακριά μπορεί να μην το έχουμε. Οπότε το δίδαγμα λοιπόν ήταν το, η δυνατότητα τη συνεργασία μεταξύ Βορρά και Νότου για να βοηθήσουμε τι χώρε υπομετάβαση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι πω έχουμε ένα πρόγραμμα στο Νότιο Σουδάν, παραδείγματο χάρη, όπου η κυβέρνηση της Νορβηγίας συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις Αιθιοπίας, της Ουγγάντα και της Κένιας για να δώσει αρρωγή στην οικοδόμηση βασικής διοίκησης σε μια χώρα που δεν είχε ποτέ τέτοια πράγματα. Οπότε άλλο ένα παράδειγμα συνεργασίας βορρά-νότου. Το δεύτερο βασικό κεφάλαιο αφορά συνεργασίες για εμπειρογνωμοσύνη και έχουμε εδώ πέρα ξεκινήσει μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να προσφέρει εμπειρία που προέρχεται από τα κράτη-μέλη και από κρατικές υπηρεσίες και από ΜΚΟ οι οποίες έχουν εμπειρία που είναι σημαντική για τη μετάβαση αυτή μετά από συγκρούσεις. Και υπ' αυτή την έννοια η διαδικασία που ξεκίνησε την πρωτοβουλία μας είχε δύο αρχές που ήταν πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά το πώς θα εντοπίσουμε αυτή την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Πρώτο ήταν ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει μόνος του αυτός ο ΟΗΕ, δεν είχαμε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη εσωτερικά το δεύτερο ήταν πως θα πρέπει να συνεργαστούμε με χώρες που έχουν εμπειρία στήριξης τέτοιας μετάβασης. Είτε ε, πρόκειτο για εσωτερική εμπειρία, είτε πρόκειτο μέσω, για εμπειρία μέσω εξωτερικών προγραμμάτων και εμπειρία που απέκτησαν έτσι. Οπότε η πλατφόρμα αυτή λέγεται CapMatch. Είναι κάτι το πολύ απλό Δηλαδή, χώρες ή αποστολές του ΟΗΕ που έχουν ζητήσει τέτοιες ικανότητες μπορεί να τις περιγράψουν με τρόπο απλό και τα κράτη-μέλη όπου οι κρατικές υπηρεσίες ή η ΜΚΟ ε, μπορούν να περιγράψουν την δική τους εμπειρία. Το σύστημα λοιπόν δίνει μετά στις χώρες την επιλογή διαφόρων πηγών εμπειρίας. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε εύκολα τις ικανότητες που χρειάζονται οι χώρες που είναι σε αυτή την κατάσταση. Το τελευταίο κομμάτι της δουλειά μας αφορά την εσωτερική μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως κάθε οργανισμός πρέπει και εμείς να δούμε τις διαδικασίες μας για να είναι αρκετά γρήγορες για να ανταποκριθούν σε αιτήματα αρρωγής από χώρες που είναι υπομετάβαση για να είναι αρκετά ευέλικτο το σύστημα για να ανταποκριθεί. Κάτι το οποίο θα τόνιζα γιατί νομίζω πως αποτελεί πρόκληση για όλους τους μεγάλους πολυμερείς οργανισμούς είναι το πώς θα συνδυάσουμε τα διαφορετικά τμήματά μας που εργάζονται στους τομείς της πολιτικής και της ασφάλειας και στον τομέα α, <clears throat> ε, της ε, ανάπτυξης. Οπότε έχουμε παραδείγματο χάρη τους συναδέλφους από τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ που εργάζονταν στο παρελθόν χωριστά όσον αφορά την στήριξη σε αστυνομία, δικαιοσύνη κτλ. Οπότε φροντίζουμε η βοήθεια αυτή να μην είναι κατακαιρματισμένη, αλλά να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε χώρες όπως η Λιβερία, η Λιβύη, η Ακτή Λεφαντοστού για να έχουμε ε, καλά αποτελέσματα. Εδώ πέρα θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Κλήφη, η οποία μίλησε πολύ λίγο, αλλά είπε πάρα πολλά, πολλά σημαντικά πρέπει να πω. Και βέβαια μπαίνουμε στον διάλογο και δίδω αμέσω τον λόγο στον κύριο Λέιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση θεωρώ πως η Επιτροπή αυτή και το Κοινοβούλιο μας αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ε, μη στρατιωτική ανοικοδόμηση χωρών και τα τελευταία χρόνια ε, είδαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς μπορεί να βοηθήσει ως μια soft power θα λέγαμε. Δεν μπορεί να την δυνατότητα στρατιωτικών ε, επιχειρήσεων αλλά βοηθάει ε, σε αυτά τα προβλήματα. Και πράγματι, ως γνωστόν, ο πόλεμος ε, γίνεται γρήγορα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η ειρήνη, ειδικά σε χώρες όπου υπάρχει, δεν υπάρχει τάξη. Και δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και λείπουν οι βασικές αυτές ικανότητες. Το ερώτημά μου είναι τι γίνεται ακριβώς όταν κινητοποιείται ο ΙΕ σε μια χώρα. Είναι μια συμφωνία με την εκάστοτε κυβέρνηση. Αν υπάρχει κυβέρνηση, πώς πάτε σε μια χώρα. Είναι μια σύμβαση με την κάθε χώρα. Μετά το ερώτημα πώς έχει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ε, είμαστε στον τομέα της ανοικοδόμησης και έχουμε διαφορές δυνατότητες μέσω της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής. Υπάρχουν καμιά φορά και ανταγωνιστικά συναισθήματα, πώς πάει η συνεργασία. Και τρίτον, είπατε πώς ενδιαφέρονται σε άλλα μέρη του κόσμου για τις εμπειρίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και ίσως στο παρελθόν Πορτογαλίας και Ισπανίας. Αλλά αν σκεφτώ τις χώρες στις οποίες αναφέρατε, δηλαδή Λιβερία, Λιβύη, Εμένη, δεν ε, μου έρχεται έτσι εύκολα τι μπορεί να διδαχτεί κανείς από μας. Είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις. Οπότε μπορούμε πραγματικά κάτι ε, από την... Ε, να διδάξουμε κάτι στις χώρες αυτές από τη μετάβαση από τον κομμουνισμό στη δημοκρατία. Να παρακαλέσω διαδικαστικά τους συναδέλφους να δοθούν όλες οι ερωτήσεις και μετά να δοθεί μια συνολική απάντηση. Η κυρία Λέζη, παρακαλώ. Ähm, Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική ανθρωπιστική αποστολή αυτή την οποία κάνετε και όλες οι χώρες στις οποίες δουλεύετε ε, πραγματικά είναι δύσκολες και είναι και πολύ περίπλοκη η δουλειά σας. Και σήμερα το θέμα μας είναι οι μη στρατιωτικέ ε, πρωτοβουλίες εγώ θα διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Λάινεν και θα έλεγα είναι πραγματικά καθαρά πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και καθόλου στρατιωτική. Και τέλος πάντων δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Θέλω να κάνω και μια παρατήρηση. Μιλήσατε κι εσείς για μια συνολική προσέγγιση με ποιον τρόπο υπάρχει σε αυτή τη συνολική προσέγγιση ε, η συνεργασία στρατιωτικής και μη στρατιωτικής πτυχής και ποια θέση έχει η στρατιωτική πτυχή. Γιατί βεβαίως ε, μας απασχολεί αυτό το θέμα είναι εδώ πέρα σήμερα και η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω εάν έχει αλλάξει κάτι εντωμεταξύ, γιατί είχαμε πολλές εμπειρίες και με την IT και υπήρχε κάτι το οποίο διάβασα ότι πριν από την τελευταία καταστροφή ούτως ή άλλως δεν ήταν πάρα πολύ καλή η κατάσταση και σύμφωνα με το παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων του ΟΗΕ το 2008 ε, ε, είχε, υπήρχε λοιμό εκεί πέρα και με 96 εκατομμύρια ε, προπολογισμό θα είχε αποφευχθεί αυτή η καταστροφή. Η, η αποστολή όμως, η Μινούστα εκεί πέρα είχε ένα προϋπολογισμό 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς το βλέπετε αυτό, πώς θα υπάρξουν κάποιε αλλαγέ στο μέλλον. Αλλά το βασικό μου ερώτημα πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση. Η εμπειρία και στο, Ιράν, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και στην ΑΙΤ έδειξε πως η μη στρατιωτική επέμβαση δεν ενισχύει και υποστηρίζει διαρκώς τις κρατικές δομές, γιατί συχνά υπάρχουν και διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά και για το ότι ε, συχνά η διαρκή στήριξη σημαίνει πως αδυνατίζουν οι δομές του ίδιου του κράτους. Και επίσης μιλήσατε για τη διαρκή οικονομική στήριξη και εκεί πέρα είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Παραδείγματος χάρη αν δούμε το Αφγανιστάν. Εκεί πέρα ξένες ε, εταιρείες ε, κάνουν τα έργα, ξένοι εργάτες παίρνουν τους μισθούς, η τοπική οικονομία δεν βοηθιέται καθόλου. Αν δούμε επίσης το Ιράκ, επίσης το τι γίνεται και εκεί πέρα νομίζω πως μπορούμε να μιλήσουμε για εδραίωση της καταστροφής. Οπότε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την, την εμπειρία ώστε οι βραχυπρόθεσμες αυτές επεμβάσεις, οι οποίες συχνά μετατρέπονται σε μακροπρόθεσμες, να λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί πέρα. Ο κύριος Ζάμπια. Ε, więc jeśli można, e, to ja przede wszystkim chciałem e, bardzo serdecznie podziękować Pani. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κλήφη για τις πληροφορίες που μας έδωσε και τώρα θα είχα μια ερώτηση ελαφρώς διαφορετική σε σχέση με τα όσα ακούσαμε. Γνωρίζουμε ότι η έξοδος από την σύραξη κάθε φορά είναι μια μακρά διαδικασία. Δηλαδή δεν σημαίνει πως επειδή αποσύρονται τα στρατεύματα τελειώνει η υπόθεση. Όμως εδώ βρισκόμαστε σε κατάσταση σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον, η έξοδος από την κρίση θα άλλα τόσα. Εδώ λοιπόν τι δυνατότητες έχουμε, ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ε, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε, ποιες είναι οι συγκεκριμένες δυνατότητες, ποιοι είναι οι ανθρώπινοι πόροι, οι ειδικοί που έχει στη διάθεσή του ΙΕ, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως είναι απαραίτητο να συνεργαστούν οι ειδικοί από διάφορους τομείς, από το νομικό μέχρι ειδικού μηχανικούς για την ε, κατασκευή του υδροδοτικού δικτύου, για παράδειγμα. Και έπειτα, οι δραστηριότητες τις οποίες εσείς προωθείτε έχουν ε, την απαραίτητη οικονομική ασφάλεια γιατί είναι δράσεις οι οποίες ε, διαρκούν χρόνια και όπου εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει κάποια σταθερότητα και κάποια εγγύηση δημοσιονομική. Και ποιος είναι ο προπολογισμό που έχει στη διάθεσή του ΟΗΕ. Οι αγορητές, οι ομιλητέ, να μου επιτρέψετε να δώσουμε τώρα τον λόγο στην κυρία Κλειφ και στη συνέχεια να περάσουμε στο δεύτερο γύρο τον συζητήσεων. Perfect. Κύριε Κλήφ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τη μεθοδολογία του ΟΗΕ και την συνεργασία μας με τις κυβερνήσεις, έχω να σας πω το εξής. Η παρουσία του ΟΗΕ στις διάφορες χώρες γίνεται με δύο τρόπους σε όλες τις χώρες παγκοσμίω υπάρχει ε, κάποια μόνιμη εκπροσώπηση από αυτές, αυτούς τους αναπτυξιακούς φορείς και υπηρεσίες μας για την μακρόπνοη αρρωγή, άρα είμαστε εκεί πέρα συνεχώς παρόντες και η μεθοδολογία μας είναι να έχουμε μια γενικότερη στατική αναπτυξιακή αιτήση των κυβερνήσεων και στη συνέχεια έχουμε ε, μια υπογραφή μια γενική συμφωνία για τις προτεραιότητες και τους τομείς που είναι επιθυμητό και βεβαίως όταν ε, ε, αυτή μας η παρουσία ε, γίνεται σε κάποιες χώρες όπου υπάρχει κάποια ξαφνική αλλαγή, μετασχηματισμός, αλλαγή, θα πρέπει να προσαρμοστούμε ταχαίως στο αυτό το οποίο κάνουμε και επίσης συνεργαζόμαστε με εκείνους ούτως ώστε να έχουμε μια ανάλυση των συγκρούσεων και έτσι να μπορούμε να είμαστε στη θέση τέλος πάντων να μπορούμε να ενεργήσουμε προληπτικά σε περίπτωση κρίση. Και ο δεύτερος τρόπος κατά τον οποίο ε, ενεργούμε ενώ όταν έχουμε την σχετική έγκριση έτοιμα της, ε, του, του, Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν υπάρχει κάποια ειρηνευτική αποστολή, κάποια διαμεσολάβηση ή κάποια σχετική πρωτοβουλία. Και αυτό σημαίνει ότι ε, αυτός ο οποίος μας στέλνει δεν είναι η κυβέρνηση βέβαια, αυτό που ζητά την παρουσία μας εκεί, είναι το Συμβούλιο Ασφαλεία. Τώρα όσον αφορά τα το, πολιτικό σκέλος θα πρέπει να υπάρχει σαφής ε, ειδική αίτηση ε, της ε, κυβερνήσεως για να μπορούμε να παρεύουμε. Το θέμα δεν είναι να παρακολουθήσουμε κάποιες εκλογές ή έστω στα τεύματα ή τελος πάντων κάποιους υπαλλήλου. Αυτό το που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε δυνατότητα στα πλαίσια κάποια κυβέρνηση, στα πλαίσια κάποια χώρα και αυτό γίνεται μόνο η αιτήση αυτή. Και έτσι μόνο είναι δυνατόν να τα καταφέρουμε. Οπότε, όσον αφορά ε, αυτό το σκέλος της αποστολής μας ε, συζητιέται, έχουν πολλές επαφές με τις κυβερνήσει για το τι είδους αρρωγή, αρρωγή θέλουν, πώς τη θέλουν και λοιπά. Επίσης έχουμε στενή συνεργασία μέσω κάποιων συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε για να σας δώσω δύο παραδείγματα. Έχουμε μία διαδικασία ανάλυσης μετά, τον, μετά τις συγκρούσεις και αυτό γίνεται στην Ιεμένη για να βοηθήσουμε την κοινωνία, να υπάρξει εθνικός διάλογος, τόσο ώστε να βάλουν, να θέσουν προτεραιότητες τους και ε, όσον αφορά τη, τον τομέα τη, της, ε, της ειρήνευσης ε, και την κοινωνία των πολιτών έχουμε μια διαρκή συνεργασία με το EIAS ούτως ώστε να μπορούμε να κινητοποιήσουμε εμπειρογνώμονες και να δούμε κάθε φορά τι θέλουμε. Αυτά γίνονται σε συνεργασία επομένω με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σημαντικά. Τώρα, όσον αφορά την συνεργασία πολιτικών στατιωτικών, ε, και αυτό είναι σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεών μας και έτσι έχουμε την, το IMPP, η, όλα, όλο αρχικά όπως ε, βλέπετε χρησιμοποιούμε full και επομένως με αυτό το μέσο ε, συνδυάζουμε τις ενέργειες των φορέων για ανθρωπιστική αρρωγή, ε, ανάπτυξη, διοκτικές αρχές, στρατιώτες κλπ. Και έτσι γίνεται ένας κεντρικός σχεδιασμός ε, και ο συντονισμός. Επίσης, πρόληψη θεομηνιών, ε, ενέργειες για την IT, όλα αυτά ήταν σε εμπειρία που χρησιμοποιείται και γενικά η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να θωρακιστεί και όχι απλώς να μαζεύει τα κομμάτια εκ των υστέρων όταν συμβεί η καταστροφή. Και τώρα μιλώ και για φυσική καταστροφή, για θεομηνία, γιατί ε, <laughs> φυσικά η ΑΕΤ ήταν πολύ πιο ευάλωτη από άλλες χώρες όσον αφορά το σεισμό, γιατί ε, τα κτίρια τα αιτινά δεν ήταν για ακριβώ φτιαγμένα για τέτοιο σεισμό, αλλά μιλούμε και για καταστροφές που προέρχονται από άνθρωπο. Δηλαδή πολέμους και συγκρούσεις. Οπότε προσπαθούμε να κατευθύνουμε εκεί όλο ένα και περισσότερους πόρους, να υπάρχει πρόληψη και έτσι να έχουν οι κοινωνίες κάποιο είδους διαμεσολάβηση εσωτερική για να αποφύγουν την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Πολλές φορές βέβαια θα προσπαθούμε να έχουμε ε, σχέση ε, κόστος αποτελέσματος καλύτερη όταν ενεργούμε των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Επίσης, ανασύνταξη, ανασυγκρότηση της οικονομίας, ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, όποτε. Γιατί αυτά πάνε χέρι-χέρι με την ε, ειδευτική διαδικασία. Γιατί αν ο κόσμος δεν έχει, <clears throat> δεν δεν δουλειά, δεν, έχει, δεν μπορεί να θρέψει την οικογένειά του, τότε πώς θα, θα αγκαλιάσουν τη δημοκρατική διαδικασία, τον δημοκρατισμό. Επομένως όλα αυτά σίγουρα είναι αναπόσπαστο τμήμα της δουλειάς που κάνουμε και φυσικά ε, όλα αυτά είναι δύσκολα και πολλές χώρες τώρα σε όλο τον κόσμο δυσκολεύονται να ε, δημιουργήσουν θέσεις εργασίας αρκετές και να χαλαρώσει κάπω το εργασιακό μέτωπο. Αλλά πάντως ε, για κάθε μετασχηματισμό αυτά είπαμε ότι είναι πάρα πολύ βασικά και πολύ σημαντικά. Οπότε τώρα ξαναγυρίζουμε στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε το ποια είναι τα συμπεράσματα, τα μαθήματα που έχουμε αντιλήσει από τις μεταβάσεις στην Ευρώπη και πόσο μπορούμε αυτά λοιπόν τα, τις εμπειρία να τη χρησιμοποιήσουμε για άλλε χώρε. Όμω, υπάρχουν διαφορέ μεταξύ ε, ε, χώρων που είχαν εμφύλιο πόλεμο και από την άλλη μεριά ε, δημοκρατικό μετασχηματισμό, χωρίς εμφύλιο από κάποιο αυταρχικό καθεστώς, αλλά πολλές φορές στην Ευρώπη αυτά τα οποία έχουν γίνει ας πούμε σχετίζονται πιο πολύ με την Τινησία και όχι τόσο ε, με την Λιβύη, γιατί στη Λιβύη ήταν πολύ πιο βίαιη η σύγκρουση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για του μετασχηματισμού που ξέρουμε, πάντα δανειζόμαστε κάποια στοιχεία και πάντα υπάρχουν και ερωτηματικά που εκκρεμούν. Α πούμε, την πρώτη φορά που πήγα στην ε, Βόρεια Αφρική μετά την Αραβική Άνοιξη, σχεδόν σε όλες τις χώρες με ρωτούσαν τι κάνετε όσον αφορά τα, τα, τους απόρριτους ε, φακέλους, τα, τα, τα μυστικά του παλαιού καθεστώτος. Να, βλέπετε τι γίνεται. Υπήρχαν εκείνα σημεία παρά τις διαφορές. Τώρα για να δούμε το τελευταίο σημείο το οποίο αφορά τη σχέση μεταξύ της δυνατότητες του ΟΗΕ και την εμπειρογνωμοσύνη μπορούμε να εισφέρουμε ε, ανθρωπιστική κρίση και έτσι προσπαθούμε να καλύψουμε τις ε, οργανώσεις να μπορούν να δρουν τομεακά για το νερό, την τροφή, υγεία, παιδεία, συνεργασία με μη κυβερνικέ οργανώσεις και στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας, την ΕΚΟ και στην περίπτωση που έχουμε ε, κάποια πολιτικές ρυθμίσεις που πολλές φορές είναι πιο εύκολο να αναπτύξει κανείς το πολιτικό προσωπικό ε, ταχαίως παρά ε, παρά όλο το οπλοστάσιο το οποίο υπάρχει από πλευρά πάλι πολιτική δράση. Ε, και θα δώσω τώρα τη σκητάλη στη Ρενάτα εδώ ε, προ τα αριστερά μου για να σα πει ακριβώ πώ κινητοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη μα. Καλημέρα σα συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ και πάλι που μας καλέσατε εδώ. Θα ήθελα να σας πω κάτι για τους πόρους και για κάποια από τα συμπεράσματα που έχει αντιλήσει ο ΙΕ είναι το ότι δεν υπάρχει μία και μόνη μέθοδος με την οποία να μπορέσουμε να, να δούμε τι γίνεται, πώς μπορούμε ταχαίως να κινητοποιήσουμε τους κατάλληλους. Γι' αυτό και εμείς έχουμε τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες και σε αυτό διαφέρουμε κάπως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα-πρώτα, ε, ε, κάνουμε ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δανειστεί από εμά ε, όσον αφορά στατιωτικέ παρεμβάσεις, αλλά αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς χρησιμοποιούμε ε, αρκετό προσωπικό για ενευτική δράση. Πάνε, πάνε, και έρχονται τέλος πάντων ε, το προσωπικό μας εκεί που χρειάζεται. Δεν εκπροσωπούμε κάποιο κράτος μέλος, δεν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο φορέα. Ε, απλό είναι αυτή είναι διεθνής υπάλληλοι. Ε, και υπάρχει φυσικά ένας μικρός πυρήνας σε κάθε αποστολή και επομένως αποστολές σε αυτούς στηριζόμαστε όπως έγινε και στην ΑΕΤ. Επίσης έχουμε το, τους ε, γρήγορους μηχανισμούς ε, κάτι το οποίο σχετίζεται με τις δυνατότητες των, ε, μελών, των κρατών ανάπτυξη δυνάμεων για ανθρωπιστική βοήθεια αλλά συγκροτούμε και τέτοιες επομένως ομάδες ε, που αυτό επίσης είναι διαφορετικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επομένως stand-by συνέχεια ε, ε, κάποια αστυνομική δύναμη και επίσης το ίδιο σχήκε για μια άλλη ομάδα, 5-6 περίπου, δικαστές, οργανιστικούς υπαλλήλους όσο αφορά τα θέματα δικαιοσύνης και αυτή η συνέχεια είναι λοιπόν stand-by όποτε χρειαστεί να παρέμβουν και επίσης αν χρειαστούμε περισσότερο προσωπικό απευθυνόμαστε στα κράτη-μέλη. Και ε, οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι κάθε φορά το τι εμπειρογνώμες χρειάζονται, τι μπορούμε να κάνουμε ε, ε, στις, στις, στις χώρες, σε επιβάση των θεσμικών οργάνων τους και γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την εμπειρία που χρειάζεται για την διακυβέρνηση της κάθε χώρας. Οπότε, εκεί πέρα πρέπει να απευθυνθούμε στο, στη χώρα για να αντιλήσουμε εμπειρία από τα κράτη-μέλη, Οπότε να συγκροτήσουμε κάθε φορά με τους μηχανισμούς που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να βρούμε το προσωπικό που χρειάζεται από την κυβέρνηση, από οπουδήποτε. Και αυτό ακριβώς είναι η ουσία του, του, του, έργου μας στα πλαίσια της σχετικής πρωτοβουλίας που έχουμε αναπτύξει. Άρα δεν υπάρχει μία και μόνη συνταγή, ένας και μόνος μηχανισμός. Να, ποια είναι η διαφορά μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σχέση με το τι κάνετε εσείς στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Έχουμε ακόμα τρεις ομιλητές, με πρώτον τον κύριο Μιλάν Μόν. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κράφη, σας ευχαριστώ. Κυρία με ευχαριστώ που ήρθατε. Η Λιβύη, όπως ξέρετε, είναι μια χώρα που αξίζει της προσοχής μας εστιάζεται λοιπόν και η προσοχή μας, είναι κοντά μας ε, και προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει όπως και προσέξαμε ε, να, να περιορίσουμε όσο γίνεται την εκατόνδη που ε, ακολούθησε την ανατροπή του Καντάφη. Για πέστε μας επομένως τι γίνεται εκεί, τι συνεργασίες υπάρχουν, γιατί από την άλλη μεριά υπάρχουν φοβερά προβλήματα ασφαλείας στη Λιβύη και είδαμε τι έγινε με αυτή την τρομοκρατική επίθεση στην ε, Βενγκάζη κατά ε, των ε, Αμερικανικών εκεί προσβευτικών προξενικών αρχών προβλήματα με τους εξοπλισμούς εκεί άρα έχουμε και το πρόγραμμα για την ενίσχυση των συνόρων και πέστε μας όμως λοιπόν δύο λόγια παραπάνω για τη Λιβύη και επίσης μια άλλη γενικότερη ερώτηση για πέστε μας το έργο σας στον ΟΗΕ πώς επηρεάζεται από την χρηματοπιστωτική κρίση, γιατί πολλά κράτη-μέλη που συνήθως σας ενισχύουν ε, εμποδίζονται, ε, δεν, δεν έχουν τους αρκετούς πόρους, ε, πάσχουν δημοσιονομικά, ας το πούμε. Για πέστε μας επομένως, πώς έχει πληγεί το έργο σας μέσα σε αυτή την κατάσταση που έχει τόσο πολύ την Δύση. Κυρία Ζακοσάρη. Kiitoksia ε, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα που μας είπατε. Λέει η κυρία Γιακονσάρη, το πρόβλημα του είναι ότι πάσα επιτυχία σας δεν προβάλλεται τόσο πολύ όσο οι ατυχείς στιγμές του έργου σας. Α, παράδειγμα, είναι το πόσα απαιτήκατε στον τελικό τιμόρ και πόσο λίγο προβλήθηκαν. Τέλο πάντων, στο θέμα του εκδημοκρατισμού, για πετε μα, πόσο πολύ πρέπει να ευαισθητοποιηθεί κανεί στα θέματα της, ε, του πολιτισμού τη κάθε χώρα, τη κουλτούρα που επικρατεί σε κάθε χώρα. Α πούμε, σε πολλέ χώρε ε, στην Αφρική η δημοκρατία λειτουργεί καλά, αλλά είναι διαφορετική δημοκρατία από αυτή που έχουμε μάθει. Ούτε το κομματικό σύστημα στις χώρες εκείνες είναι το ίδιο με το, αυτό που έχουμε στην Ευρώπη. Άρα, για πετε μας εσείς, πώς προετοιμάζεστε, τι στάση, τι συμπεριφορά τηρείτε όσον αφορά αυτούς τους δημοκρατικούς μετασχηματισμούς αυτής της χώρας, πώς προσαρμόζεστε τις ανάγκες κάθε χώρας. Thank you, Mr. I also want to thank you and it is already a good tradition. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πιστεύω πως είναι μια ήδη πολύ καλή παράδοση αυτή που δημιουργούμε εδώ να καλούμε τον γενικό, την Γενική Γραμματέα του ΙΕ. Πάμε στην Νέα Υόρκη εξάλλου σύντομα και ίσως θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε εκεί αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω γιατί η ανταλλαγή απόψεων ήδη δείχνει, αν πάμε σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ότι πρέπει να συζητήσουμε τα προβλήματα ή τις ε, προκλήσεις. Εγώ πιστεύω ότι όταν πάμε σε μια χώρα, στην ουσία πάμε για να στηρίξουμε την ε, χώρα να ανακάμψει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο του συστήματος του ΙΕ. Και εδώ μιλάμε για τη συνεργασία με την Ένωση. Όμως, πιθανότατα δεν είναι τόσο εύκολο αν λάβουμε υπόψη τη γενική συζήτηση στην Γενική Συνέλευση και ενώ εξετάζουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση μιας χώρας, ε, το πώς θα παρέμβουμε και πώς θα στηρίξουμε τη διαδικασία συμφιλίωσης ε, και σε ποιες περιφέρειες της χώρας. Ε, αν είναι, ας πούμε, καλό στην Αφρική, στη Σομαλία κτλ θα πήγαινε προσωπικό από τη ΣΥΠΑ, ως εμπειρογνώμονες, ως ε, δομές σε πλατφόρμες που μπορούν να στηρίξουν ε, την ενίσχυση του κρατικού συστήματος της χώρας. Αν πάμε σε άλλες περιοχές, ίσως είναι, είναι πιο προβληματικό. Πώς λοιπόν εξισορροπείται η αναζήτηση εμπειρογνωμόνων που πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη διαρκή ε, οικοδόμηση των πολιτικών δομών, ε, των δομών των κοινωνικών σε κάποια χώρα. Δεύτερον, πρέπει να συνδεθούν οι δικές σας δραστηριότητες με την γενικότερη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οπότε, Πιστεύω πως κάποιες φορές ε, το θέμα αυτό είναι πολύ λεπτό. Και έπειτα, ποια είναι η πείρα σας ε, από τη συνεργασία με την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε συγγνώμη, με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εσείς συνεργάζεστε στην ποινική δίωξη και στην αναζήτηση των ε, ε, εγκληματιών και ποια χρήση κάνετε των δομών για τις οποίες μόλις μιλήσαμε. Ευχαριστώ. Μεγάλη χαρά έχω που σε βλέπω Σάρα και στη συγκεκριμένη θέση γιατί ξέρω πόσες ικανότητες και εμπειρία έχεις. Να δεν ξεχνάμε τη σπουδαία έκθεση που συνέταξες για το UNDP ακριβώς για τη σημασία του κράτους δικαίου στις αναπτυξιακές πολιτικές. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω Αναπτύσσοντας τα όσα είπε, ε, σας ρώτησε ο συνάδελφος Μίλαρμον για τη Λιβύη. Μήπως θα μπορούσατε να μιλήσετε και για την μεταβατική δικαιοσύνη στην ε, Λιβύη. Δεν είναι μόνο το θέμα της ασφάλειας, αλλά και της ε, δικαιοσύνης. Ο ΙΕ και μάλιστα πρόσφατα έστειλε έναν ε, εξαίρετο εκπρόσωπο στη Λιβύη, τον Ιαν Μάρτιν, αλλά αυτά τα θέματα ξεπερνούν το Διεθνές Δικαστήριο. Και, και, και το την ανάμειξή του σε όλες αυτές τις δίκες πιθανότατα θα ασχοληθεί με τις δίκες των πιο σημαντικών, των πιο γνωστών ανθρώπων στην περιοχή. Αλλά υπάρχουν χιλιάδες κόσμος, κυρίως νέοι άνδρες από τις γειτονικέ χώρες που, που τόσκασαν απλά από τις φυλακές στην Τρίπολη. Και δεν υπάρχουν οι δομές για κάτι τέτοιο. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς το παρακολουθείτε αυτό. Και έπειτα το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν κανείς δεν μιλά πια γι' αυτό. Λες και ξαφνικά ε, ε, έχει τελειώσει η μεταβατική περίοδος εκεί και φυσικά βλέπουμε ότι η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο ε, με το ρόλο των Αμερικανικών δυνάμεων. Μπορεί όντως ο ΙΕ να χρειάζεται να παρέμβει και να ενισχύσει και η δικαιοσύνη εκεί μεταξύ, άλλων, μεταξύ πολλών άλλων είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και επίση εκεί πρέπει να, κατασκευαστούν οι κρατικέ δομέ. Ποια είναι τα σχέδια για το Αφγανιστάν από πλευρά του ΙΕ Και τέλο, αναπτυσσόμενη χώρα. <coughs> όπου υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίες διότι μόλις πέθανε ο δικτάτορα εκεί, η Αιθιοπία. Είναι μια χώρα όπου πιστεύω ο ΙΕ κατάλαβε τι παίζεται, αλλά δεν έκανε και πολλά, γιατί βέβαια είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκούσαν λάθος πολιτική, παριστάνοντας ότι ο δικτάτορας ε, ήταν ένας αξιοσέβαστος, ε, ε, μια αξιοσέβαστη προσωπικότητα, δεσμευμένη και προσιλωμένη στην ανάπτυξη. Τώρα όμως βλέπουμε ότι γίνεται χαμός. Έχουν, ε, ε, έχουν εφημώσει τον τύπο. Βλέπουμε εντάσεις ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς που ποτέ δεν υπήρχαν. Τώρα ξαφνικά ανακύπτουν γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί όντως να παρέμβει στον διορισμό των μουσουλμάνων ε, ηγετών. Επίσης γίνεται ε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για βασικά θέματα του κράτους δικαίου και είναι μια χώρα που θεωρητικά είναι σε μετάβαση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το ρόλο του ΟΗΕ εκεί και την εξέλιξη αυτού και την ε, συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο τον έχετε σημαντικά ερωτήματα, αναμένουμε σημαντική απάντηση. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι, για τις εξαιρετικές ερωτήσεις που θέσατε. Θα ξεκινήσω με τα ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατάσταση σε κάθε χώρα και ίσως και μετά με πιο γενικ... θα, θα ασχοληθώ με τα γενικότερα θέματα πολιτικής. Όσον αφορά τη Λιβύη, όπως γνωρίζετε, Τη στιγμή όπου η διεθνή κοινότητα μπόρεσε να παρέμβει, ε, συνέχισαν να ε, επιμένουν τα πολιτικά, τα προβλήματα ασφαλείας και οι πολιτικές διαδικασίες ήταν πολύ πρώιμες, στα πολύ πρώιμα στάδια για την ε, δημιουργία μιας κυβέρνησης που θα είχε την νομιμότητα τοπικά ώστε να μπορεί να λάβει κάποιες αποφάσεις για θέματα προτεραιότητας. Είναι μια δύσκολη περίοδος όσον αφορά τη διεθνή βοήθεια γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει υπάρχει ε, προθυμία να σταλεί βοήθεια, αλλά όχι πάντοτε για στήριξη της πολιτικής διαδικασίας τοπικά. Ε, εκεί ε, νομίζω ότι αυτό τώρα αλλάζει, πιστεύουμε ότι αλλάζει αυτό, έχουμε την επιβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι το κάνει αυτό. Καταρχήν θα πρέπει εκείνοι να θεσπίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητές τους και μετά να δημιουργηθούν κάποια βασικά υπουργεία που δεν υπήρξαν ποτέ πριν ε, σε μια φυσιολογική σχέση με τους πολίτες. Μια πρώτη περίοδος λοιπόν θα είναι αυτό το βασικό επίπεδο δημιουργίας θεσμών και οι λιβικές αρχές έχουν ζητήσει βοήθεια για τη δημιουργία κάποιων από αυτών των βασικών κυβερνητικών λειτουργιών. Αναμένουμε πως η στήριξη στην πολιτική διαδικασία θα εξακολουθήσει να είναι προτεραιότητα και ότι τελικά θα υπάρξει και ένα αίτημα για στήριξη στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καθώς και με την οικονομική αναζωγόνηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Έχει ζητηθεί βοήθεια για την εκμάθηση πρακτικών προσεγγίσεων όσον αφορά την ε, ε, την ε, συμμετοχή των δύο φίλων ε, στην πολιτική και στη δικαιοσύνη. Επίσης ζήτησαν βοήθεια για μεταβατική δικαιοσύνη και φυσικά θα πρέπει να σας τιμήσουμε για το ρόλο που παίξατε στο Ανατολικό Τιμόρ. Ε, το θέμα της μεταβατικής δικαιοσύνης στη Λιβύη αλλά και στις άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι στο επίκεντρο των ετοιμάτων για αλλαγή. Είναι ένα από τα πράγματα που είδαμε να γίνεται ο μεγαλύτερος θόρυβος από τον κόσμο ε, σταδιακά γίνεται κατανοητό ότι οι μεταβατικές ε, διαδικασίες αυτού του τύπου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε 6 μήνες ή ένα χρόνο για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν διότι πρέπει ε, να, να συλλεχθούν πληροφορίες, να γίνουν έρευνες και να γίνουν και διώξεις, οι οποίες διαδικασίες παίρνουν όλες χρόνο, αλλά και η μεταβατική δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Συμπεριλαμβάνεται δημιουργία μιας κοινωνικής συνένεσης για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και η διάχυση αυτής της συνένεσης από μηχανισμούς όπως η δημόσια επικοινωνία, ε, σύστημα ενημέρωσης κτλ. Ακόμα λοιπόν και σε αυτές τις χώρες που, θεωρούμε ότι κάναμε καθολική δουλειά και ότι έχουμε κάνει ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταβατική δικαιοσύνη στην Χιλή για παράδειγμα διέρχεσε 20 με 25 χρόνια αυτή η διαδικασία και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Είναι θέμα προτεραιότητας λοιπόν. Μπορούν να γίνουν πράγματα για να ξεκινήσει σωστά η διαδικασία. Το μήνυμα ε, είναι ότι θα είναι μακρά η διαδικασία και ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Και αυτό θα βοηθήσει ολόκληρη την ε, περιοχή. Να ε, μιλήσει για το Αφγανιστάν η Ρενάτα και μετά θα επανέλθω στις γενικότερες ερωτήσεις περί πολιτικής. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι αναφέρατε ότι το Αφγανιστάν έχει ξεχαστεί για την ώρα. Είναι μια ξεχασμένη σύγκρουση και είναι εντυπωσιακό για όσους από εμά έχουμε δουλέψει εκεί και δεδομένων των προκλήσεων που υπάρχουν. Είναι ένα παράδειγμα για μεταβα... μεταβατικών οροσίμων. Όταν λέμε μετάβαση, σημαίνει ότι ο δυτικός κόσμος αποσύρει τις δυνάμεις του και τις διεθνείς δυνάμεις της ΣΥΣΑΦ. Όμως η μετάβαση στο Αφγανιστάν περιλαμβάνει διάφορα σημεία. Ε, ένα βασικό ορόσημο θα είναι οι εκλογές που θα γίνουν το 2014. Είναι ένα παράδειγμα για το πας ε, δυναμική είναι μια διαδικασία μετάβασης και ένα παράδειγμα για το πώς ε, η προσοχή μπορεί να αποσπαστεί ιδιαίτερα όσον αφορά δημοσιονομικούς περιορισμούς και δυσκολίες Πολλοί κόσμος ε, θα είχε φανταστεί ότι ο, ο νόμος του ΟΗΕ ε, θα είχε αρθεί από, τον... Ε, από τη στιγμή που αποσύρονται οι διεθνείς δυνάμεις. Οι Αυγανοί όμως δεν σκέφτονται κάτι τέτοιο. Ε, γιατί καθώς οι χώρες αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν οι αναπτυξιακές ενισχύσεις και οι συμβολές προς τον ΟΗΕ και είναι πραγματικά ηρωνικό το ότι η ΟΝΑΜΑ κλείνει τώρα 10 γραφεία σε ολόκληρο το Αφγανιστάν που ορισμένα είναι μικρά καθώς αποσύρεται η ΆΙΣΑΦ. Αυτά είναι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι. Ένα-δυο σημεία που έχω να πω για το Αφγανιστάν είναι, και εσεί μιλήσατε για την τοπική οικονομία και τη σημασία αυτής, δεν θέλουμε απλώς να βρούμε πώς θα βρούμε βιώσιμους ε, τρόπους για να ε, τροφοδοτήσουμε την οικονομική αναβίωση, αλλά πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο της παρουσίας μας. Η τοπική οικονομία έχει αλλάξει, έχει μεταλλαχθεί λόγω της παρουσίας των διεθνών δυνάμεων και μάλιστα με την ε, απόσυρση της διεθνούς παρουσίας υπάρχει μια ολόκληρη τοπική βιομηχανία που θα καταρρεύσει όλοι αυτοί που προσφέρουν υπηρεσίες στις στρατιωτικές βάσεις, αυτοί που μεταφέρουν ε, ε, διάφορα προϊόντα, τοπικοί συνεργάτες κτλ. Πρόσφατα είδα αποτελέσματα, στηρίζονται 9 με 15 Αφγανοί από αυτόν που εργάζεται και συνεργάζεται με τις στρατιωτικές βάσεις. Θα είναι ένα σημαντικό θέμα. Μια προτεραιότητα λοιπόν είναι πώς θα διατηρηθεί η διεθνής δέσμευση εκεί. Και μια από τις προτεραιότητες του ΟΗΕ είναι αυτή ακριβώς. Πώς θα διατηρηθεί η δέσμευση μετά από την απόσυρση από εκεί. Η δέσμευση πολιτική, οι ανθρώπινα δικαιώματα και εστιασμός στην... στην ε, ε, δημιουργία κυβερνητικών θεσμών. Ε, να μπορέσουμε δηλαδή να διευκολύνουμε τους Αφγανούς, να τους στηρίξουμε. Πώς το κάνουμε αυτό, πώς εξισορροπούμε τις σχέσεις με πιο ισότιμο και βιώσιμο τρόπο. Γιατί κάποιες φορές ε, ξεχνάμε πόση πρόοδο έχουν σημειώσει οι Αφγανοί. Μετά από τρεις δεκαετίες αδελφοκτόνων πολέμων έχουν ε, πολύ καλή διαχείριση ας πούμε των οικονομικών τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλά χρήματα που περνούν από τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Έχουν ένα μεγάλο ποσοστό επίσης συμμορφωμένων ανθρώπων που ξεκινάνε όμως από μια βάση όπου το 70% του κόσμου ήταν αναλφάβητο μετά από τρεις δεκαετίες πολέμου. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν το, το, το μέγεθος της πρόκλησης. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τη φύση της διεθνούς ε, ε, δέσμευσης. Τα Βαλκάνια είναι μια, ένα καλό παράδειγμα. Πώς ε, δηλαδή διατηρείς μια σχέση από τη στιγμή που αλλάζεις τον ίδιο τον ιστό και το Αφγανιστάν θα είναι πρόκληση. Όταν ε, ε, βέβαια και η απόσυρση των ε, δυνάμων ασφάλειας θα είναι ένα θέμα κλειδί. Σας ευχαριστώ. Και έρχομαι σε κάποια άλλα ερωτήματα για το τι διδάγματα αποκαμίσαμε από τις προσεγγίσεις μας και από την πολιτική μας. Καταρχήν για τη δημοκρατία και τις επαφές και τα μοντέλα τα οποία προβάλλουμε. Πάντοτε είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε την περιοχή του εκδημοκρατισμού νομίζω ότι πέρα από την γενική συνένεση επί της αρχής πολύ λίγο πειραματισμός έχει γίνει με διάφορα μοντέλα συμμετοχής. Συχνά λοιπόν θεωρούμε ότι είναι οι ηγέτες αυτοί που προκύπτουν από τις εκλογές και δεν έχει γίνει πολλή δουλειά για το ποιες είναι οι υπόλοιπε δημοκρατικές πρακτικές και μηχανισμοί που ταιριάζουν στις κοινωνίες ανάλογα με τους καιρούς. Ω τμήμα λοιπόν αυτής της πλατφόρμας για την οποία μίλησα προσπαθούμε να ε, συλλέξουμε εμπειρίε από διάφορες χώρες, από διάφορα είδη δημοκρατική συμμετοχή που βρήκαν πως ήταν αποτελεσματικά σε μεταβατικές περιόδους και ω ένα παράδειγμα που είναι πολύ ανορθόδοξο και ένα μη φυσιολογικό τρόπος. Η Μποτζουάνα, για παράδειγμα, περιέγραψε το παραδοσιακό τη σύστημα και μετά του μηχανισμού που χρησιμοποίησε ώστε να έχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση νέων και γυναικών μέσα στο ίδιο σύστημα. Εμείς θεωρούμε πως είναι καλό ότι δηλαδή να καταλάβουμε πως οι αρχές είναι παρόμοιες και να ενθαρρύνουμε την κοινοτομία με βάση διάφορους μηχανισμούς συμμετοχής. Κάτι άλλο το οποίο έχει προκύψει και στη συζητήση της ΣΥΦΚΑΤ για τα διάφορα μοντέλα δημοκρατικής εκπροσώπησης ήταν η σύνδεση ανάμεσα στη δημοκρατία και την ακραία φτώχεια, ανέχεια ή ανισότητα. Χρειάζονται επιπλέον έλεγχοι κάποιες φορές για να παρεμποδιστεί ε, η χειραγώγηση της δημοκρατικής διαδικασίας όταν υπάρχει μια διαδικασία εκδημοκρατισμού σε ε, συνθήκες εξαιρετικής ε, φτώχειας ή ανισότητας. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για την εξορρόπηση της πρόσβασης των κρατών μελών όσον αφορά την συμμετοχή και την παροχή εμπειρογνωμόνων με την αποδοχή διαφόρων εμπειρογνωμών από διάφορες χώρες προέλευσης και σε διαφορετικές καταστάσεις. Είναι σαφές στις διαδικασίες του ΟΗΕ ότι πάντοτε το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο απευθυνόμαστε στα κράτη-μέλη για να ζητήσουμε οτιδήποτε. Αυτό είναι προϋπόθεση. Δεν υποδεικνύουμε καμιά προτίμηση για κάποιο κράτο μέλος. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις ε, υποδοχής ε, μπορούν να ζητήσουν δική επιγνωμοσύνη. Ε, κοιτούν, ας πούμε, χώρες που υπήρξαν παρόμοιες εμπειρίες και όντως τους ευθαρρύνουμε να το κάνουν αυτό. Γιάννη, προσπαθούμε να εξορροπήσουμε την γνώση της γλώσσας και των ε, ε, τοπικών εθινόντων και παραγόντων με την ε, δυνατότητα και την εμπειρία παρόμοιων καταστάσεων, γιατί πιστεύουμε ότι η συνεργασία ανάμεσα στις βόρειες και τις νότιες χώρες στην παροχή βοήθειας ε, ε, δεν έχει, δεν έχει εξεπιθεί αρκετά. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα παροχής βοήθειας από κάποιες χώρες της Ένωσης, αλλά είναι ε, σπάνια τα παραδείγματα. Θα πρέπει ίσως να το διερευνήσουμε, πως είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε πιο συστηματικά, γιατί υπάρχει δυνατότητα να συνδυάσει όλη την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση θεσμών, συνδυασμένες με κάποια τοπικά, τοπικές δυνατότητες ή ικανότητες, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να διαβιβαστούν αυτές οι εμπειρίες. Επίσης έχει να κάνει με την μακρά παράδοση της, ε, ε, της Ένωσης ε, για τη δημιουργία θεσμών με αραβικές χώρες, χώρες και τα κτλ. Ευχαριστώ. Παραγωγική συζήτηση και είχαμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Γκλή και τους συνεργάτες της που αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο του σήμερα να είναι κοντά μας. Ευχαριστώ.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 Ladies and gentlemen, we are going... Κυρίες και κύριοι, λέει ο πρόεδρος, να συνεχίσουμε την συνεδρίασή μας. Και τώρα θα πάμε στο ρυθμό 4 σημείο της διάταξης, που είναι η έκθεση προόδου σχετικά με την Αλβανία για το 2012. Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση ε, της ε, εκθέσεως για την ε, Αλβανία, που είναι η πρώτη-πρώτη σε μια σειρά ψηφισμάτων που αφορούν τις χώρε των μελουσών διευρύνσεων. Όπω γνωρίζετε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα και πρότεινε να χορηγηθεί, να απονεμηθεί τέλο πάντων το καθεστώ τη υποψηφία προσέγγιση χώρα στην Αλβανία, ε, επιφυλασσομένων βέβαια των όσων προβλέπονται από τη Συμφωνία για τις μεταρρυθμίσει σε κοινοβούλιο, δικαιοσύνη κλπ. Τώρα, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Χουντή. Ο κύριος Χουντής είναι ο εισηγητής μας ο οποίο πρόκειται να μα εξηγήσει τι δικέ του θέσει όσον αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Χουντή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Όπως εξήγησε ο Προεδρεύων της Επιτροπής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, είναι η πρώτη συζήτηση της έκθεσης προόδου, ενταξιακής προόδου για την Αλβανία και να συμπληρώσω ότι η Επιτροπή, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δουλεύουμε με το χρονοδιάγραμμα το ψήφισμα το σχετικό να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας και με αυτό βαδίζουμε. Ε, θέλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι την έκθεση την έχετε μπροστά σας. Ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις επισκέφθηκα την Αλβανία στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι η δεύτερη επίσκεψη από τη στιγμή που ανέλαβα τη σχετική ευθύνη. Σε αυτή την επίσκεψη την τελευταία συναντήθηκα με όλους τους πολιτιακούς και πολιτικούς παράγοντες, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της κυβέρνησης, όλα τα πολιτικά κοινοβουλευτικά κόμματα της Αλβανίας, συνδικαλιστικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ε, επίσης, ε, ε, συνεργασία με την Αλβανική Πρεσβεία των Βρυξελών. Γιατί το λέω αυτά. Θέλω να τους ευχαριστήσω διότι οι συζητήσεις ήταν ειλικρινείς και η εικόνα που μου έδωσαν έδειχνε την πρόθεση, την επιθυμία για να αποκτήσει η Αλβανία το ενταξιακό καθεστώς και ταυτόχρονα μπορώ να πω την επιθυμία να δουλέψουν ακόμα περισσότερο προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι όροι. Με αυτή την έννοια λοιπόν τους ευχαριστώ πολύ και οι σχετικές παρατηρήσεις έχουν πάρει υπόψη το υλικό, τα στοιχεία και τις συζητήσεις αυτές. Δεύτερο, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν, διότι και με την Κομισιόν και τους ε, υπεύθυνους ε, συνεργαστήκαμε. Ε, η έκθεση της, όπως είπε ο Προεδρεύων, η έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τη διεύρυνση που παρουσίασε πρόσφατα ο κύριος Φούλε και οι επιμέρους παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα της Αλβανίας με βρίσκουν σύμφωνο, έχουν ληφθεί υπόψη όσο αφορά τη δική μας την έκθεση και ιδιαίτερα σχετικά με τα βήματα που έχουν γίνει για τις 12 προτεραιότητες και επομένως έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη και στη δική μας την πρόταση. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέβαλε σημαντικά και βοηθάει στη συγκρότηση αυτής της έκθεσης. Παίρνω κατευθείαν στο πιο ουσιαστικό θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μην σας κουράζω με τα επιμέρους θέματα, τα οποία δεν θεωρώ ε, δευτερεύοντα βεβαίως. Σχετικά με το καθεστώς απόδοσης υποψήφιας χώρας στην Αλβανία. Η πρόταση την οποία διατυπώνω, που στο σχετικό σημείο προτίθεμαι να την κάνω πιο καθαρή και πιο σαφή, με σχετική τροπολογία, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει, συμφωνεί να δοθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας στην Αλβανία, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Εδώ θα ήθελα τη γνώμη σας, τη γνώμη και των μελών της Επιτροπής, ούτω ώστε να έχουμε, έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε ομόφωνοι σε αυτό το βασικό ζήτημα α, και παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι με, ένα, με μια τέτοια εισήγηση, μια τέτοια πρόταση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δίνει ένα σήμα προς την αλβανικέ αλβανικές πολιτικές δυνάμεις και στον αλβανικό λαό θα δίνει μια ενθάρρυνση να συνεχίσουν αυτές τις προσπάθειες και θα επισημαίνει και ποιες κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι οι προσπάθειες που πρέπει να συνεχιστούν. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι, επειδή θα είμαστε ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε εκλεγμένο θεσμό πρέπει οι δικές μας επισημάνσεις και παρατηρήσει, παρατηρήσεις, και αυτό κάνει η δική μου έκθεση, να έχει έντονο το κριτήριο ότι όλα αυτά, όλη αυτή η προσπάθεια, οι μεταρρυθμίσεις, τα προβλήματα που υπάρχουν θα πρέπει να αποβλέπουν καταρχήν και εν τέλει θα έλεγα στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, στη βελτίωση από άποψη δικαιωμάτων τη ζωή του λαού τη Αλβανία και των πολιτών τη Αλβανία. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι στο σχετικό θέμα που τοποθετούμε ε, πολύ συγκεκριμένα που είναι το κεντρικό, νομίζω ότι το ψήφισμά μας, θα ακούσω και τους άλλους συζητητές, θα πρέπει να έχει σαφέστατη την πρόθεσή μας, την πρότασή μας να αποκτήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας, βάζοντας βεβαίως α, την ε, επισημένοντας με συγκεκριμένο τρόπο το τι ακόμα πρέπει να γίνει. Εκεί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, γιατί νομίζω ότι πρέπει να υποθεί αυτό διότι όπως θυμόσαστε ε, αγαπητοί συνάδελφοι το κεντρικό πρόβλημα που είχαμε στην προηγούμενη αξιολόγηση της ε, πορείας και της κατάστασης της Αλβανίας ήταν το πολιτικό πρόβλημα. Από την εικόνα, από την ενημέρωση και από αυτά που ξέρουμε όλοι φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Δεν ξέρω αν έχει σταθεροποιηθεί, αλλά φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Έχει προχωρήσει η συνένεση στην αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων. Είναι σημαντικό ότι σε αυτή την προσπάθεια υποβοηθούν και άλλε πολιτικέ δυνάμει, όχι μόνο οι δύο μεγάλε πολιτικέ δυνάμει. Εν πάση περιπτώσει, Εφόσον αυτό το πολιτικό κλίμα έχει βελτιωθεί, η συνένεση, η συμφωνία στο να λυθούν προβλήματα ή να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες για έναν καλύτερο κανονισμό, λέω παραδείγματος χάρη στη Βουλή, ε, της, της Βουλής, για την, ε, το θέμα της ασυλίας και το χτύπημα της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο. Και στα άλλα θέματα νομίζω ότι είναι μια καλή προϋπόθεση ε, για να πούμε ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια με καλύτερες ε, όρους και να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτό είναι ένας βασικός λόγος που ε, η πρόθεσή μου, η πρότασή μου είναι το ψήφισμά μας να έχει αυτή την ε, τοποθέτηση, δηλαδή να δοθεί στην Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Τώρα, δύο κουβέντες για τα υπόλοιπα, για να μην σας κουράζω περισσότερο. <clears throat> Στο, στο σχέδιο του ψηφίσματος, στο σχέδιο της έκθεσης, έχετε φαντάζομαι δει τα θέματα που αναφέρονται. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι η περιορισμένη αρχική έκταση που μπορεί να έχει αυτό το ψήφισμα δεν, τα έχει, δεν έχει όλα τα σημεία που θα ήθελα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Ε, έχει τα βασικά, μπορούμε να τα συμπληρώσουμε και εννοώ ότι με τροπολογίες και δικέ μου και φαντάζομαι περιμένω να ακούσω σχετικέ τροπολογίε, να γίνουν σχετικέ επισημάνσει, ούτω ώστε το ψήφισμα και το περιεχόμενό του να ολοκληρωθεί στο τι ακριβώ πρέπει να γίνει. Γενικά, αν μου ζητάτε μια εικόνα, ε, ε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να γίνουν. Θα επισήμενα περισσότερο τα θέματα που έχουν σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Ε, δεν, δεν, δεν, δεν υποτιμώ την ανάγκη του να ενισχυθεί και να εξηγενθεί το δικαστικό σύστημα, το θέμα της διαφθοράς, το θέμα ε, εν γέννη του κράτους δικαίου, αλλά ε, κατά τη γνώμη μου η επισήμανση έχει το χαρακτήρα περισσότερο ε, να παρθούν μέτρα, να βελτιωθεί η κατάσταση των πιο αδύναμων, κατά τη γνώμη μου, κοινωνικών στρωμάτων και εκεί οπωσδήποτε το σχετικό, η, σχετική πρότασή μου δίνει μια έμφαση, το ομολογώ. Ε, επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό ότι με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε και με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή γενικώ, ε, θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε ως θετική τη στάση της Αλβανία στη σχέση με τις γειτονικέ χώρες και εδώ νομίζω είναι σημαντικό αυτή η όθηση που θέλει να δώσει το ψήφισμά μας να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ την ε, στάση αυτής της Αλβανία σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η περιοχή των Βαλκανίων και που σωστά και με αυτό τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είπατε με τη σημερινή έκθεση ξεκινάμε τη διαδικασία του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει, α, ακούσαμε και την Κομισιόν, τι θα γίνει με την υπόθεση τη ένταξη, μάλλον ή του καθεστώτο ή τη ένταξη των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Επομένω, το μήνυμα που θα εκπέμψουμε σχετικά με την Αλβανία θα έχει και μια ευρύτερη επίδραση και, στην, ε, και στις άλλες χώρες και θέλω να πιστεύω ότι το, ε, η Επιτροπή μας και τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει το σωστό μήνυμα ότι οι χώρε αυτές, η, η προοπτική τους είναι να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκεί να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις σε όφελος του λαού τους του και των πολιτών τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χούντι. Ξεκινάει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στον διακεκριμένο συνάδελφο τον ε, κύριο Λίμπο Ρότζεκ, σκιώδη ηγητή από του Σοσιαλδημοκράτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να συγχωρούμε τον κύριο Χούντι για την έκθεσή του. Είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω δίνει το σωστό πολιτικό στίγμα, τονίζει τα θετικά, αναφέρει και κάποιες αδυναμίες που έχει ακόμα η Αλβανία και μιλάμε για τη θετική πτυχή, ναι, η έκθεση αναγνωρίζει την πρόοδο της Αλβανίας το τελευταίο έτος και τονίζει πως η πρόοδος αυτή έγινε λόγω της συνεργασίας των ε, μεγαλύτερων πολιτικών δυνάμεων στην κυβέρνηση και βεβαίω στην αντιπολίτευση. Όσον αφορά τα προβλήματα, κάποια από τα επίμονα προβλήματα, κράτος δικαίου, δημόσια διοίκηση, ο αγώνας κατά της διαφθοράς κτλ. Οπότε, να τονίσω και πάλι, το βασικό πολιτικό μας μήνυμα πρέπει να είναι πως απαιτείται μια εσωτερική συνένεση, μια σχέση επίσης λειτουργική μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, να εδραιωθεί η δημοκρατία στην Αλβανία και βεβαίως η, το βασικό είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας. Οπότε υποστηρίζουμε πλήρως τη γραμμή του ΣΥΤΗ, αλλά βεβαίως θέλουμε να ενισχυθούν κάποια σημεία στην έκθεση, όπως παραδείγματο χάρη η διατύπωση στην παράγραφο 124, που πρέπει να είναι πιο έντονη η διατύπωση για να φανεί η πλήρης στήριξη της πρότασης της Κομισιόν για να δοθεί ε, στην Αλβανία το καθεστώς ε, της υποσχείας χώρας ε, υπό όρους βεβαίως. Δεδομένου του ότι δεν είχαμε πέρυσι έκθεση για την Αλβανία, Νομίζω πως θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην σημασία της ε, συμφωνίας ε, του Νοεμβρίου 2011 που έδωσε τέλος στην πολιτική στασιμότητα και επέτρεψε πορεία προς τις 12 προτεραιότητες. Επίσης σημαντικό είναι η εκλογή, ε, η εκλογή του διαμεσολαβητή που μπορεί επίσης να αναφερθεί στην έκθεση. Είναι σημαντικό αυτό για την ενίσχυση της αλβανικής δημοκρατίας και την ενθάρρυνση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό το οποίο θα έχει σημασία στην Αλβανία του χρόνου θα είναι οι εαρινές ε, βουλευτικές εκλογές. Αυτό πρέπει να, όχι μόνο να αναφερθεί, αλλά και να τονιστεί νομίζω στην έκθεση. Είναι δηλαδή σημαντικό και για την ανάπτυξη της αλβανικής δημοκρατίας, αλλά θα αποτελέσει και τη λιδία λίθο για την πρόοδο της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εγγυηθεί δηλαδή το καθεστώς υποψηφίας χώρας. Ο κύριος Χουντής επίσης αναφέρθηκε για, κάποια, για τα ασθενέστερα τμήματα της αλβανικής κοινωνίας, είτε είναι οι φτωχοί, ανέφερε τους, ε, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Εγώ θα αναφέρω και τα δικαιώματα των παιδιών που είναι επίσης πρόβλημα στην Αλβανία. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό στην έκθεση επίσης. Πρέπει να αναφέρουμε πως η Αλβανία δεν έχει ακόμα ακυρώσει το καθεστώς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Νομίζω καλό είναι να υπέθυμίσουμε στις αλβανικές αρχές να το κάνουν. Και τέλος, να αναφέρω τα ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Η Αλβανία τα τελευταία χρόνια έχει παίξει πολύ θετικό ρόλο. Πρέπει νομίζω να το αναγνωρίσουμε αυτό ναι, εντονότερα. Παράδειγμα του χάρη να δούμε τι γινόταν στη, στη γειτονική Πουγουδουμού. Ε, η Αλβανία έπαιξε επικοδομητικό ρόλο στο να ηρεμήσουν τα πνεύματα και οι εντάσεις. Και ελπίζω η χώρα να συνεχίσει σε αυτή τη γραμμή. Συνοψίζοντας λοιπόν η να πάρα πολύ καλή, ναι, έχουμε λίγες τροπολογίες, αλλά νομίζω πως θα έχουμε καλές αθαρρυντικές εκθέσεις και επικοδομητικά επίσης τονίζουμε κάποια από τα σημεία σε κάποιους τομείς όπου η Αλβανία ε, έχει ακόμα δουλειά μπροστά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Σχάκε που είναι πιο δυσυγήτρια για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Νομίζω πως ε, μπορούμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά στο σημαντικό αυτό θέμα. Είναι σημαντική αρχή, αλλά είναι η αρχή μιας μακράς ή εντατικής διαδικασίας μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να είναι βαθιές και όχι επιφανειακές. Το Κοινοβούλιο έχει δει από πρώτο χέρι την πολιτική πόλωση που ακόμα υφίσταται στο πολιτικό σύστημα της Αλβανίας και πρέπει να συνεχίζουμε να μιλάμε και να απευθυνόμαστε απευθεία στο λαό της Αλβανίας. Αυτό το κάνουμε για το καλό τους και όχι για μια πολιτική τάξη ή γενιά. Και ελπίζω ο αλβανικός λαός και όλες οι πλευρές του πολιτικού φάσματος να συνεργαστούν επικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας θεωρήσουν ε, ε, ε, έναν διαμεσολαβητή. Το έλεγα και στο παρελθόν και το γνωρίζει βέβαια, και ο πρόεδρος. Συνολικά λοιπόν δεν μετράει μόνο και το αποτέλεσμα, αλλά και η διαδικασία που θα ακολουθεί είναι εξίσου σημαντική και πρέπει να έχει νόημα και να συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Κάποια πράγματα που είναι σημαντικά για εμάς. Πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε από εδώ και μπρος όλες οι διαδικασίες και χώρες ένταξης να, έχουν, να δίνουν περισσότερο βάρος στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι σημαντικό. Τα κεφάλαια 23 και 24 θα ανοίγουν πρώτα και θα κλείνουν τελευταία. Αυτό θα είναι λοιπόν σημαντικό πλαίσιο για τις συζητήσεις μας για μεταρρυθμίσεις στα σημαντικά ζητήματα αυτά στο μέλλον. Καλωσορίζουμε επίσης το δόγμα της μηδενικής ανοχής για συστημικά προβλήματα διαφθοράς που πρέπει να γίνει για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις δημόσιους θεσμούς και βέβαια είναι προαπαιτούμενο για δημοκρατική μεταρρύθμιση, αλλά βεβαίω όταν μιλάμε για μηδενική ανοχή πρέπει να υπάρχουν και δίκαιες δίκες και σωστές διαδικασίες. Δεν μπορεί να είναι μονομερή η διαδικασία η καταπολέμηση της ατιμορρησίας είναι πάρα πολύ σημαντική, είτε μιλάμε για διαφθορά, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή γενικώ. Τρίτον, για αυτούς που εξαρτώνται από το κράτος, οι άνθρωποι στις φυλακές, παιδιά στα αρφανοτροφία, ε, οι πνευματικά ασθενείς. Πρέπει οι συνθήκες τους να βελτιωθούν συστηματικά. Όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, θέλουμε να τονίσουμε τα εγγυημένα δικαιώματα για τους ΛΟΑΤ και τους ΡΟΜΑ και τις λοιπές μειονότητες. Είναι σημαντικά αυτά. Τέλος, πλουραλισμός στα ΜΜΕ, ελευθερία στα ΜΜΕ και ψηφιακή ελευθερία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ομάδα μας και μάλλον θα υποβάλουμε τροπολογίες ε, όπως περίπου τις ανέπτυξα και αναμένουμε την συνεργασία έτσι ώστε αυτά τα οποία λέμε ως μεταρρυθμίσεις να μεταφραστούν σε κάτι το οποίο θα νιώσει ε, ο αλβανικός λαός πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα με την άδειά σας θα μιλήσω εγώ ως ε, πρόεδρος αντιπροσωπείας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη να σας ενημερώσω πως ε, θα αλλάξω πολλές ιδιότητες κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να καλωσορίσω την έκθεση αυτή, καθώς έχει περάσει πολύ καιρό από όταν υιοθετήσαμε το προηγούμενο ψήφισμα για την Αλβανία. Σύμφωνο με τους προλαλήσαντες πως ο κύριος Χουντής ε, προετοίμασε μια πολύ καλή έκθεση αλλά θεωρώ πως είναι καθηκόν μας να την κάνουμε ακόμη καλύτερη με το να καταθέσουμε τροπολογίες για να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει συγκεκριμένα την Αλβανία στα περαιτέρω βήματά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά η Αλβανία παλεύει εδώ και καιρό με εσωτερικά πολιτικά προβλήματα τα οποία αποτελούσαν τροχοπέδι και καθυστερούσαν την πρόοδο της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω να σημειώνεται πρόοδος στο να ξεπερνώνται αυτά τα εμπόδια και στο να ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος ειδικά για βασικά ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη. Αυτό αναμέναμε από τους Αλβανούς πολιτικούς εδώ και καιρό. Επίσης, είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Το καθεστώς υποψήφιας χώρας για την Αλβανία είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά εξαρτάται από την πολιτική βούληση και τον σταθερό πολιτικό διάλογο μεταξύ όλων των δυνάμεων του πολιτικού φάσματος. το να πω πως θέλω να είμαι αισιόδοξο είναι ισοπροβολικό. Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξο και να δω την περαιτέρω πρόοδο και ομαλοποίηση της εσωτερικής πολιτικής ζωής στη χώρα. Ελπίζω επίσης πως οι προσεχείς εκλογές δεν θα ανακόψουν αυτή την πρόοδο. Όσον αφορά την έκθεση, σύμφωνο πλήρως με τον εισηγητή πως πρέπει να ενθαρρύνουμε τους Αλβανούς πολιτικούς να συνεχίσουν τον πολιτικό διάλογο και να γίνει αυτός ο διάλογος βιώσιμος και μόνιμος. Μόνο έτσι θα εκπληρωθούν οι υπόλοιπες προτεραιότητες τις οποίες ανέφερε η Κομισιόν ως κλειδί για την περαιτέρω διαδικασία ενοποίησης. Εξυπακούεται πως οι νόμοι για το ανώτο δικαστήριο, την δημόσια υπηρεσία μαζί με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου πρέπει επίσης να εγκριθούν. Όμως δεν είναι μόνο η έγκριση των νόμων. Η Αλβανία πρέπει να εφαρμόσει αυτούς τους νόμους και να αποκτήσει και ουσιαστική εφαρμογή τους, ειδικά στις προτεραιότητες ε, που αναφέρει η Κομισιόν. Μόνο τότε θα μιλήσουμε για απτή πρόοδο. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω δύο συγκεκριμένους τομείς που πρέπει να εξτάσουμε πιο λεπτομερώς στην έκθεση. Το πρώτο αφορά την δικαιοσύνη, κατά πολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι σαφές πως η αιστεία σημασία αυτών των τομέα είναι κέρια σημασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως η Αλβανία θα είναι προετοιμασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η ανεξαρτησία και η ελευθερία των ΜΜΕ εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και θα παρακολουθώ στενά το θέμα αυτό στο πλαίσιο και της έκθεσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Κοπά από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον συνάδελφο Νίκο Χουντή για την έκθεσή του για την Αλβανία που νομίζω καλύπτει όλα τα βασικά σημεία σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της χώρας. Ε, θέλω και εγώ να πω ότι είναι πολύ θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων το γεγονός ότι η Αλβανία σημείωσε πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και ε, κατάφερε να εκπληρώσει αρκετά από τα κριτήρια ένταξης. Πρέπει λοιπόν να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή εισηγείται την απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει αυτή την εισήγηση υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι είναι μόνο η αρχή ενός μακρύου δρόμου που προϋποθέτει εντατικοποίηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Μερικές σύντομες επενσημάνσεις. Πρώτα απ' όλα η εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας, ένας ε, τομέας όπου εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια πολλά προβλήματα, ε, η εύρυθμη λοιπόν λειτουργία του Κοινοβουλίου πρέπει να αποτελεί τον κανόνα από εδώ και πέρα και δεν πρέπει να επιτραπούν πισωγυρίσματα. Μεγαλύτερες προσπάθειες απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της δικαιοσύνης, τη διαφθορά, καθώς επίσης και την προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Σε σχέση με το θλιβερό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες επαγρύπνησης και ενημέρωσης των γυναικών για τα δικαιώματά τους, καθώς και να αναπτυχθεί το δίκαιο υποδοχής κακοποιημένων γυναικών και των οργανισμών παροχής συμβουλευτικής στήριξης στα θύματα κυκλωμάτων διακίνησης γυναικών και παιδιών. Αναφορά στην κατάσταση στις φυλακές και στις περιπτώσεις κακομεταχείρισης κρατουμένων υπάρχει ήδη στο προσχέδιο της έκθεσης. Πρέπει πάντως να εκφράσουμε την ανησυχία μας και για την απαράδεκτη πρακτική προφυλάξης ανηλίκων για μεγάλες χρονικές περιόδους. Καθήκον της δικαιοσύνης είναι να προστατεύει το συμφέρον των παιδιών, και είναι δύσκολο να κατανοήσω πώς η μεταχείρισή τους ως εγκληματίες, πριν καλά-καλά εκδικαστεί η υπόθεσή τους, μπορεί να εξυπηρετεί το συμφέρον αυτών των παιδιών και του συνόλου της κοινωνίας. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Αλβανία, κάτι το οποίο τονίζουμε για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η Αλβανία πρέπει γρήγορα να υιοθετήσει την απαραίτητη νομοθεσία για την αποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων και να ολοκληρώσει την απογραφή του πληθυσμού σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κοπά. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οφείλω να σας πω ότι με χαροποιεί το να συζητούμε για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Αλβανία με μια συζήτηση επικοδομητική και ανυφάλια. Πρέπει να μας χαροποιούν τέτοια μαντάτα γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με την Αλβανία. Έχουμε εξαιρετικό εισηγητή στην πολιτική μας ομάδα. Ε, η εισηγήτριά μας τέλος πάντων ε, έχει πάρα πολλές γνώσεις και παρακολουθεί την πορεία της εξελίξης στη χώρα, Οπότε, το θέμα είναι ότι έχουμε κυβέρνηση και αντιπολίτευση που έχουν βρει ε, έναν κοινό τόπο τόσο ώστε να μπορέσουν να διεξάγουν έναν νυφάλιο διάλογο ε, τουλάχιστον όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτή επομένω είναι μια αλλαγή προς το καλύτερο που έλαβε χώρα. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές που θα διεξαχθούν. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό να πούμε στην Αλβανία ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το, αυτή τη γραμμή πλεύση. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή μας ε, η ουδέτερη θέση όσον αφορά την προσέγγιση της χώρας. Νομίζω στο παρελθόν ήμασταν κάπως προκατηλημένοι, ας το πούμε κάπως υποκειμενικοί ε, και είχαμε κάποιες πολιτικές ομάδες που υποστήριζαν τις δικές τους δυνάμεις. Ήταν πιο επίοικείς με τους πολιτικούς τους εκεί συμμάχους και ήταν πιο αυστηροί με τις υπόλοιπε πολιτικέ δυνάμει στη χώρα. Πάντως, το μήνυμα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το μήνυμα που είναι να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν έχουμε εδώ, δεν παρίσταται κάποιο συνεργό από του πράσινου και πρέπει να επισημάνουμε ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε ότι σοβεί στην Αλβανία από τι επισκέψει μα εκεί. Ότι θα πρέπει να δούμε τι επιδόσει τη χώρα όσον αφορά το περιβάλλον και ότι γίνεται όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τι γίνεται με τον τουρισμό. Θεωρώ ότι ε, αυτού του είδου η παράδοση του να ε, προσέχει στο περιβάλλον είναι μια παράδοση που δεν την έχει η Αλβανία, δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το μέτωπο και συμφωνώ με αυτούς που μίλησαν για τον ε, δημιουργικό ρόλο της Αλβανίας όσον αφορά την γενικότερη γεωπολιτική της περιοχής. Τι να σας πω, πριν από τρεις μέρες στο, στα γήπεδα πάντως μας, νίκησε η Αλβανία. Τα γήπεδα πάντως οι περισσότεροι από του παίκτε Αλβανία που μα νικήσαν τι προάλλε γεννήθηκαν στο Κωσυφοπαίδιο. Μήπω θα πρέπει η Αλβανία να παίζει με δικού του παίκτε και όχι με δανεικού από το Κόσοβο. Thank you very much. Uh, I would uh, πάρα πολύ και τώρα. Θα απευθυνθώ στον κύριο Μαραγκό που είναι πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα παρουσιάσει όσο μπορεί πιο σύντομα τι θέσει του. Thank you, Mr. Good morning to everybody. Κύριε Κούκαν, σας ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Από πλευρά μου σας ευχαριστώ τα εξής. Στο παρελθόν η συνεργασία μας με τις αλβανικές αρχές ήταν πάρα πολύ αγαστή και όχι μόνο με τις αρχές, αλλά τα πήγαν πάρα πολύ καλά και με τα άλλα κρατικά όργανα και τους άλλους θεσμούς της χώρας, τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ε, όπως τις μη κυβερνικές οργανώσεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί σχετιόταν με την ε, πετυχημένη συνεργασία που συνεχίστηκε και φέτος. Είναι επομένως σημαντικό να συνεχίσουν ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτή τη συνεργασία. Φυσικά να έχουμε ενιαία φωνή, έτσι να στέλνουμε το μήνυμά μας προς τους Αλβανούς φίλους σε σχέση με την ευρωπαϊκή του πορεία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συμβολή όσον αφορά τι ε, αλλαγέ που να γίνουν στη χώρα. Πάντως, το βασικό θέμα αναφέρθηκε και η Κομισιόν το λέει στην εκθεσή τη Είναι αυτή η συνένεση που έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι έχει αποδώσει αποτελέσματα φέτος. Υπάρχει δεδομένη πολιτική συμφωνία που υλοποιεί αυτή την συνένεση και είδαμε και κάποιες αλλαγές πολύ συγκεκριμένε και σημαντικές, κάποιες που εκκρεμούσαν πολλά χρόνια. επιτέλου ολοκληρώθηκαν και χρειάστηκαν συμβιβασμοί από όλες τις πλευρές. Ασυλίε, εκλογικός νόμος κλπ. Αναφέρουμε στην εκθεσή μα και άλλα θέματα Πέρασαν όλα τα νομοσχέδια που εκκρεμούσαν, διαμεσολαβητής, διαδικασίες λήψης απόφασης από διάφορα θεσμικά όργανα και άλλα, άλλα συγκεκριμένα διαβήματα που γίνανε σε σχέση με το κράτος δικαίου. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη μέθοδο, η Αλβανία θα πρέπει να κινηθεί προς ε, την εκπλήρωση των προποθέσεων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να τι απονείμουμε το καθεστώ τη υποψηφία χώρα. Αλλά θα πρέπει να δει και τι άλλε προτεραιότητε που εκκρεμούν. Αυτά όλα που ανέφεραν οι προλαλήσαντε και άλλα. Θα πρέπει τα κριτήρια τη Κοπενχάγης να πληρώνται και κυρίω τα πολιτικά κριτήρια. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξουν οι πραγματεύσει. Γι' αυτό σα λέω. Θεωρούμε ότι τον μπαλάκι στο γήπεδο και της Αλβανίας αλλά και εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τι προσπάθειε αυτέ. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τις επιδόσεις τη η χώρα. Έχουμε τις προποθέσει που έχουμε τάξει εμείς που είναι πολύ συγκεκριμένε. Και ε, απαιτούνται κάποιε συγκεκριμένε προσπάθειες πρόοδο και στον πολιτικό διάλογο, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται να υπάρχει κάποια συνέχεια όσον αφορά τις ε, προσπάθειες σε όλους τους άλλου τομεί, αυτού που έχουμε μνημονεύσει στην ε, έκθεσή μας και νομίζω ότι και εδώ το είπαν πολλοί από τους ε, αγωγητές. Επίσης, να σας τονίσω ότι είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα της χώρας να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την ίδια δέσμευση όσον αφορά το γραμμένο έγκλημα, την καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, με, με δυναμικές έρευνες για της οδού και έτσι να υπάρχει εξασφάλιση, βεβαιότητα προ όλε τι κατευθύνσει και κυρίω προ το λαό τη χώρα ότι δεν υπάρχει ατιμορρησία όσον αφορά την εγκληματικότητα. Εμεί θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τι προσπάθειε αυτέ και χέρι-χέρι με εσά μετράμε ποντάρουμε στη βοήθειά σα τόσο ώστε η Αλβανία να μπορέσει να σημειώσει βήματα πρόοδου στην Ευρωπαϊκή Ρότα. Ε, εκεί χρειάζονται επίση πόροι και, και πολιτικοί και τεχνική, τεχνοκρατική, να συνεχιστεί αυτό ο διάλογο. Νομίζω ότι αυτή όλη η προβληματική είναι πολύ σημαντική για να αποκτήσει κίνητρο η χώρα, να δει ότι είναι ανοιχτό ο ευρωπαϊκό δρόμο άπαξ και πληρούνται τα κριτήρια αυτά τα οποία έχουμε τάξει. Thank you, Mr. Maragos. There are no more... Ευχαριστούμε κύριε Μαραγκέ. Δεν έχουμε άλλα να ζητούν το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χουντή αν θέλει να κάνει κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις ε, παρατηρήσεις και τις ε, συμπληρώσεις και τις βελτιώσεις που έκαναν προφορικά και με τις τροπολογίες. Σπέβδω να δηλώσω ότι ο εισηγητής δεν έχει κανέναν εγωισμό, ότι λέει το καλύτερο ή τα είπε όλα και επομένως θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε ούτως ώστε η έκθεσή μας, στο τελικό ψήφισμα, γίνει το καλύτερο δυνατό. Γιατί το λέω αυτό και δεν θα σας κουράσω. Γιατί είναι εύκολο, αγαπητοί συνάδελφοι, να φτιάξει μια έκθεση καλή, κακή και να λες αυτό πρέπει να κάνετε, το άλλο πρέπει να κάνετε. Η δυσκολία βρίσκεται σε αυτόν που παίρνει το μήνυμα και που πρέπει να δείξει τη βούληση ότι θέλει να τα κάνει για δικό του καλό, όχι γιατί το λέμε εμείς. Παρόλα αυτά, το μήνυμα που εκπέμπουμε ήδη από σήμερα, καθώς βλέπετε ότι η συνεδρίασή μας καλύπτεται κυρίως από αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι όλες οι πολιτικές ομάδες, αυτό κατάλαβα κύριε Πρόεδρε, της Επιτροπής μας, στα βασικά συμφωνούμε. Και επομένως εκφράζουμε μια κοινή θέληση του Ευρωκοινοβουλίου, λέω κατ' επέκταση, να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια του αλβανικού λαού, επισημένοντας με τρόπο που θέλουμε να βοηθήσουμε, ξαναλέω, ποια προβλήματα πρέπει να λύσουν. Να το πω αντιστρόφω, ε, η έκθεσή μα που θα γίνει καλύτερη να μην εκλειφθεί ω μάθημα αλλά ω επισημάνσει αναγκαίε προκειμένου να υπάρξουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τον αλβανικό λαό. Και η δεύτερη μου παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, είναι πράγματι το κρίσιμο θέμα που μα έκανε όλου να είμαστε θετικοί πια στην υποψηφιότητα είναι ότι έχουμε βήματα στο θέμα της συνένεσης κυρίως κυβέρνηση και αντιπολίτευση το να αντιμετωπίσουν με δημοκρατικό τρόπο ορισμένα θέματα. Αυτό είναι πράγματι το κρίσιμο σημείο που δεν το είχαμε σε προηγούμενε περιόδους. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτό πρέπει να σταθεροποιηθεί. Η συμφωνία του Νοεμβρίου δοκιμάζεται κατά καιρού όσο αφορά την εφαρμογή της και την ε, απόδοση αποτελεσμάτων. Σωστά επισημάνθηκε ότι μπροστά υπάρχει και η δοκιμασία από την άποψη τη διαδικασία και τη πολιτική βούληση, όχι των αποτελεσμάτων των εκλογών. Στι προηγούμενε περιπτώσει είχαμε τι πρώτε εκλογέ, τι δεύτερε εκλογέ και εκεί τα πράγματα οξύνονταν. Είχαμε μια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να δούμε πώ μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Εύχομαι λοιπόν το μήνυμα που θα εκπέμψουμε και που εκπέμπει ε, και ελπίζω να είναι και απόφαση του Συμβουλίου προ τι ε, αλβανικέ πολιτικέ δυνάμει να, ε, να εκλειφθεί με τη σωστή διάσταση του θέματος και να μην ξαναπάμε σε καταστάσεις αβεβαιότητας, μη συνένεσης, θα έλεγα μη διαλόγου, πολιτικού διαλόγου. Επομένως, οι κανόνες του δημοκρατικού διαλόγου που πρέπει να εμπεδοθούν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να, από τη δική μας την πλευρά να επισημαίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν θα επεκταθώ στα άλλα θέματα γιατί θα δω και τι τροπολογίε. Το γενικό πνεύμα δεν έχω, ξαναλέω, να συνεργαστούμε μπορεί να γίνει προφανώ καλύτερη η έκθεση και να είμαστε πιο εύστοχοι στι παρατηρήσει μα. Και σα ευχαριστώ εκ των προτέρων για τι τροπολογίε και για τι παρατηρήσει που έγιναν και που θα. μια συλλογική προσπάθεια να το τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και να δώσουμε το καλύτερο μήνυμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά, έτσι τώρα ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σας θυμίσω πως η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 22 Οκτωβρίου στις 18, 6 δηλαδή το απόγευμα. Το σημείο 5 έχει αναβληθεί όπως συμφωνήσαμε, οπότε τώρα θα δούμε την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και τη δημοκρατία και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Ο κύριος Ντόνσκης είναι ο εισηγητής και πρόκειται για την πρώτη φορά που συζητάμε στην Επιτροπή μας την ε, έκθεση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2011 μαζί με τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει οι ευρωβουλευτές. Ε, θέλουμε να υιοθετηθεί το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια που είναι αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα με την ε, επίδοση του βραβείου Ζαχάροφ. Η προετοιμασία λοιπόν για αυτή την ε, έκθεση είναι αρκετά εντατική. Όπως και παλιότερα η ετήσια μας έκθεση ανταποκρίνεται στη ε, ε, έκθεση της Ένωσης ε, για το 2011 αλλά είναι και μια ευκαιρία για τον καθαρισμό των θέση και των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου για τις ευρωπαϊκές πολιτικές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν να δώσω το, το, ε, το λόγο στον εισηγητή, κύριε Ντόνσκης, να σας θυμίσω ότι η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί στη συνεδρίασή μας στις 6 Νοεμβρίου. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση εδώ στην ΑΦΕΤ. Θα ήθελα να μοιράσω την, την σύντομη παρουσίαση σε τρία τμήματα. Καταρχήν να σας πω περί πρόκειται, δεύτερον δυσκολίες και προκλήσεις και τρίτη ε, τμήμα κάποιες επεξηγηματικές παρατηρήσεις. Θα πρέπει να σας ομολογήσω κύριε Πρόεδρε ότι ε, είχα μια τάση να ακούγομαι πολύ ακαδημαϊκός και αποσπασμένος γιατί η φιλοδοξία μου και στόχος μου ήταν και είναι ακόμα να έχουμε ένα χρήσιμο και πρακτικό έγγραφο αλλά όχι έναν κατάλογο περίπλοκο κατάλογο πρακτικών και προβλημάτων. Γι' αυτό πιστεύω πως είναι σημαντικό να έχουμε ένα πολύ στοχευμένο και χρήσιμο έγγραφο, χρήσιμη ετήσια έκθεση και γι' αυτό το λόγο η φιλοδοξία μου είναι να σχηματίσουμε το μέλλον ε, και όχι απλά να αντικατοπτρίσουμε τα στοιχεία του παρελθόντος ή του παρόντος, να έχουμε έναν αντίκτυπο στα άλλα θεσμικά ε, κοινοτικά όργανα και ελπίζω και σε τρίτες χώρες. Με χαρά λοιπόν σας λέω ότι Έχουμε κοινό έδαφο, οι συνάδελφοι και εγώ εύκολα συμφωνούμε για τα πιο θεμελιώδη ε, θέματα που αφορούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παραβίασή του σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε και τη σωστή διατύπωση. και κάποιες φορές να ξαναδουλέψουμε κάποιο υλικό ή την πρακτική πτυχή του λόγου μας. Γι' αυτό και το πνεύμα της συλλογικότητας είναι πολύ σημαντικό για μένα ε, γιατί χρειάζεται κάποια ευελιξία και χώρος ε, ελιγμού ώστε να μην ε, χαθούν τα θέματα μεγάλης σημασίας. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους λοιπόν για την υποβολή των σχολείων τους. Δεύτερο θέμα, δυσκολίες και προκλήσεις που πρέπει να τις ε, παραδεχτώ, η, η ελευθερία θρησκείας και πίστης. Εδώ νομίζω πως θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας. Δεν θα πρέπει να είναι ένας μακρύς και επαναληπτικός κατάλογος θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα ή πίστη, πράγμα το οποίο δυστυχώς προέκυψε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πω το εξή σημαντικό. Θα πρέπει να εξηγήσω γιατί αναφέρεται η Κίνα και η Ρωσία στην έκθεση. αναφέρεται γιατί αυτές οι δύο χώρες αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το φάσμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραβιάζουν ε, ε, ε, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι δύο τεράστια κράτη σημαντικά κράτη που καλύπτουν ένα τεράστιο έδαφος ε, απάτριδων πολιτισμών, μειονοτήτων, ε, θρησκευτικών, κοινοτικών, ε, ένα σωρό, και ένα σωρό ήδη μειονότητες που ζουν εκεί. Και δεν μπορώ πάνω να σας αναφέρω τον Λούσιαν Πά, έναν Αμερικανό-Κινέζο ιστορικό, που, που είπε ότι η Κίνα είναι ένας πολιτισμός ένας πολιτισμός μοιρασμένο σε ένα τεράστιο κράτος, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη Ρωσία. Όσον αφορά το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παραβιάζονται εκεί. Φυσικά συζητώντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις δεν μπορώ να παρακάμψω ένα πολύ σημαντικό τομέα τους συναδέλφους χωρίς τον οποίο τη συμβολή δεν ε, θα μπορούσα να ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και ευχαριστώ τους, ε, την Ρενάτε Βέμπερ, τους ε, υπόλοιπους συναδέλφους των Φιλελευθέρων, την κυρία Κιλ Νίλσεν και τους Πράσινους, την κυρία Άννα Γκόνες, την κυρία Βερζιά τον κύριο Γιώργο Λάιτφριτ, την κυρία Άννα Ζαπόρσκα, τον κύριο Τόκε, την κυρία Αντρικένα, για να σας πω μόνο μερικούς από τους συναδέλφους που έκαναν πολύ σημαντικέ προσθήκες και κατέθεσαν πολύ ε, ευφυεί τροπολογίε. Και τέλος κάποιες επεξηγηματικές παρατηρήσεις, ε, κύριε Πρόεδρε, για να αποφύγουμε την επικάλυψη και την επαναληπτικότητα, προσπάθησα να αντισταθώ στην πρόκληση να προσαρμόσω μάλλον να, ε, ενσωματώσω όλες τις τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Το στυλ, κάποιες ενοποιητικές αρχές, η σαφήνεια, η συνοχή ήταν αυτά που επικράτησαν. Δεν ήθελα να αποφύγουμε ένα κατάλογο δεδομένων ε, σκέψεων. Νομίζω ότι ως προς την ουσία έχουμε ε, κοινή βάση κοινό έδαφος δεν υπήρξαν διαφωνίες είτε ε, απορίες, ε, μόνο με κάποιες διαφορές διατύπωσης. Ε, οι στυλ, οι συνάδελφοι μου έδωσαν μου έδωσαν τα πιο σημαντικά στοιχεία της πολιτικής ζωής, δηλαδή τις, ε, τις κριτικές τους και την ανταπόκρισή τους. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στόκης δεν είναι εδώ, αλλά μου ζήτησε να σας παρουσιάσω τις παρατηρήσεις του για τη συζήτηση αυτή και αυτό θα πράξω αμέσως. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό χαιρετίζει το ότιος η έκθεση ξεκαθαρίζει ότι θα πρόκειται για ένα στρατηγικό έγγραφο για το μέλλον μας με προοπτική της μελλοντικέ εξελίξεις και γι' αυτό το λόγο είναι επίσκαλο δεχούμενες οι τροπολογίες που θα είναι συμβατές με το ότι θέλει συστηματικά, ε, εντατικά και εξαντλητικά να γίνεται η διαβούλευση αυτή με, το, με την Αντιπροεδρία και θα πρέπει να έχουμε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. θα πρέπει όμως να συνεχιστεί η συνεργασία με την εξωτερική υπηρεσία, ακριβώ όπω είχαμε ως προηγούμενο και σε σχέση με την ευρωπαϊκή Άνοιξη. Θα πρέπει σκεφτεί η ελευθερία να κατοχυρωθεί παντού στον κόσμο, να έχουμε μόνο τροπολογίε, γιατί υπάρχουν ενισχυτικά μαντάτα από αυτό το, το μέτωπο, όπω α πούμε τι γίνεται στο Θιβέτ, και άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε προ συμβαστικέ τροπολογίε. Είμαστε περί τροπολογία, ώστε να υπάρχουν κάποιε κοινοτικέ ε, κατευθυντήριε γραμμέ για την ε, θρησκευτική, για την θρησκεία ε, τη κυρία Αντρικένη, α πούμε, του 377, και θα πρέπει επομένω να συνεργαστεί ε, το Κοινοβούλιο με την κοινωνία των πολιτών. Επίσης δεν μπορούν παρά να χαιρετήσουν το ότι η Συρία, η Λιβύη και η Λευκορωσία αναφέρονται συχνά πυκνά στην έκθεση και ότι θα πρέπει σε αυτά τα σημεία να σημειωθούν συμβαστικές ε, τροπολογίες. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κάποιο είδους ε, αποστολές παρατηρητών για εκλογές και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε συμβασμούς για τις ρήτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές συμφωνίες. Σας ευχαριστώ και τώρα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοπά. Thank you. Uh, my colleague Lightfried cannot, uh, who is the shadow, could not be here, so I will read his presentation. Dear colleagues, you... Σας ευχαριστώ. Αναπληρώνω βεβαίω την ισχυρή συγκεκριά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρωπινά δικαιώματα και εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε την πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν έχουν υπάρξει βελτιώσεις και τι πρέπει ακόμα να γίνει. Επίσης θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να επισημάνω ακόμη μια φορά την σημασία του ορισμού του ειδικού αυσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνολικά 404 τροπολογίες έχουν κατατεθεί η έκθεση του κ. Είναι μια καλή βάση, αλλά κάποια πράγματα λείπουν. Πέντε τομεί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για εμένα. Πρώτον, η ευρωπαϊκή πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εμένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο μέλλον η Ένωση να μιλάει με μία φωνή και βεβαίως να έχει στεναρή στάση όσον αφορά τις ε, παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πρέπει να βαθμίσουμε λοιπόν ε, το έργο αυτό και να αποκτήσει την ίδια σημασία με ζητήματα οικονομικά. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι πρώτοι και όχι αγορές δεύτερον ανθρώπινα δικαιώματα και εμπόριο. Ω μέλο τη Επιτροπή ΙΝΤΕ έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα στην έκθεση αυτή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι πολυμερεί συμφωνίε για να προωθήσουμε δικαιώματα όπω η ελευθερία του συνέρχεσθε, του συνεταιρίζεσθε, η κατάργηση της παιδικής εργασίας και των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας. Ε, επίσης, η εταιρική κοινωνική ευθύνη στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου θα προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί ιδιαίτερα. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω όσον αφορά την Κολομβία, την σημασία της προστασίας των συνδικάτων και των δικαιωμάτων τους, ε, το δικαίωμα του συνέρχεστε, πρόσβαση υπηρεσίες κτλ. Τρίτον, αραβική άνοιξη και η προστασία των βλόγερ, δημοσιογράφων κτλ. Παρακολουθήσαμε όλοι τις δραστηριότητες κάποιων αρχηγών ε, κρατών όπως ε, της Αιγύπτου, Συρίας, Λιβύης κτλ. Βρένουν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που μάχονται για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία γνώμης. Γι' αυτό θέλω να καταθέσω μία τροπολογία για να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος εξαγωγών ειδικά αντικειμένων διπλής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικών αρχών και ελευθερίας λόγου. Επίσης σημαντικές ε, τεχνολογίες υποκλοπών και παρακολούθησης ε, κινητών ε, τηλεφώνων και στοχευμένης παρακολούθησης της χρήσης του ίντερνετ. Τέταρτον, δικαιώματα γυναικών και παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί στενά με τον ΟΗΕ και με οργανισμούς σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τα δικαιώματα των γυναικών. Επίσης κατέθεσα μια τροπολογία για το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην υποσαχάρια Αφρική για το ότι παιδιά κατηγορούνται για μαγεία με σοβαρές συνέπειες από τον εξωστρακισμό μέχρι τη δολοφονία τους καθώς και τις τελετουργικές θυσίες παιδιών. Πέμπτον, διακρίσεις. Ανησυχούμε για τα γεγονότα θρησκευτικής ε, μη ανεκτικότητας και βίας. Γι' αυτό ζητάμε από τα κρατημέλη να σταματήσουν τις διακρίσεις με κάθε αφορμή. Φύλλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό και διάφορα πιστεύω. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ε, διασκευτικοί διάλογοι σε διάφορα επίπεδα είμαι αισιόδοξη πως θα βρεθεί ένας καλός συμβασμός μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Το σημαντικότερο είναι να εστιάσουμε στην προστασία των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εντό και εκτό τη Ευρώπη. Τέλο, θα ήθελα να αναφέρω πω η έκθεση αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Κοπά. Κυρία Γκόμε. Πρώτα πρώτα να σας συγχαρώ γιατί αυτή η έκθεση είναι εξαιρετική και νομίζω ότι εδώ πριτανεύει το συναλληλικό πνεύμα και η κυρία Κοπά ήδη τοποθετήθηκε εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη Πότε θα ήθελα να πω πέραν της συμφωνίας μου μετά όσα ακούσαμε, να σταθούμε επομένω σε δύο-τρία σημεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι αιτήσει εκθέσεις στο μέλλον θα λαμβάνουν υπόψη το πόσο έχει λάβει υπόψη η υπάτη εκπρόσωπος της εκθέσεις μας. Και βεβαίως θα πρέπει να εμπλέκεται και ο κύριος Σταύρος Λαμπρινίδης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και επομένως ε, οι αιτήσεις έκθεσης να καλύπτουν και αυτή την πτυχή. Η επιτυχία πάσης στρατηγικής εξαρτάται από το πώς συνδυάζεται, πώς συναρθρώνονται οι προσπάθειες των θεσμικών οργάνων. Το κοινοβούλιο δηλαδή θα πρέπει να, να, να εξασφαλίζει τη συνεργασία της υποπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Ακριβώς όπως αναφέρθηκε. Έχει σημασία και το εμπόριο, η ίντα, η βιομηχανία. Ε, οι σχέσεις επομένως των επιμέρους πολιτικών που ασκούμε αντικατοπτρίζονται στην αξιοπιστία μας για το τι θα γίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό και ο ρόλος βέβαια της υπάρξης εκπροσώπου έχει βέβαια διπλό ρόλο και αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι συμπτωματικό. Ακριβώς αυτό γίνεται ούτως ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί μια τέτοια συνεργασία, ένα συντονισμός. Και αυτό πρέπει να υπάρχει συντονισμός και με το Συμβούλιο. Και φυσικά να διαπνέουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλες τις τομεικέ πολιτικές της Ένωσης. Επίσης, είναι κατακλείδη. Δεν μπορώ να συμφωνήσω 100% με την έκθεση του κ. Ντόνσκης όσον αφορά την πάγια πρακτική οι, οι χώρες, οι ομάδες χωρών να θέλουν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Δικαιωμάτων, αλλά προσοχή. Αυτό αποτελεί πάγια πρακτική. Και όμως είναι πάρα πολύ επιβλαβές όσον αφορά την αξιοπιστία αλλά και την ε, ε αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε, πρέπει να σταθεί στο επίπεδό του προσοχή επομένω στι προσπάθειε που γίνονται να αλλάξει αυτή η τάση. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήβο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο που είναι στην πολιτική μας ομάδα, τον κύριο Ντόνσκης. Είναι πολύ ε, ευαίσθητη η προσέγγιση την οποία επέλεξε για να συντάξει αυτή την έκθεση. Το θέμα είναι δύσκολο. Και δυσκολία να βρει κανείς την ισορροπία μεταξύ του συγκεκριμένου αλλά και του να έχει και μια σφαιρική προσέγγιση ταυτόχρονα. Ενώ δεν αποκλίνει από τις θεμελιώδεις αξίες. Πάντως, είναι σαφές ότι ο εισηγητής θέλησε να εστιαστεί περισσότερο σε αυτές τις γενικές αξίες και αρχές, να μην επισέλθει στις λεπτομέρειες. Οι δε τροπολογίες, όπως και η δική μου τροπολογία, αφορούν τις, ε, τα, τα συγκεκριμένα καυτά προβλήματα. Κατονομάζουμε προβλήματα και τις χώρες όπου αυτά υπάρχουν. Να επομένω η αναγκαιότητα της ισορροπίας. Τελικά επομένω θα έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις δικές μας ανησυχίες για πρακτικές, για κακές πρακτικές σε ορισμένε χώρες. Σημαντικό πάντως σε αυτή τη φάση είναι το πώς οι εκθέσεις αυτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα πώς θα περιέχουν και, κάποιες, κάποια πολιτικά μηνύματα. Κάθε μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται σημαντική ε, δήλωση πολιτική. Όπως ας πούμε έχουμε και κάποια άλλη έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι αμερικανική ας πούμε που αφορά τις πρακτικές που ισχύουν παγκοσμίω. Άρα όπως και οι Αμερικανοί και εμείς να γίνουμε πρωταγωνιστές σε αυτή τη σκηνή. Και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε την αξιοπιστία μας αλλά και έτσι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκοσμία σκηνή και να είμαστε επομένω ανεκτικοί όσον αφορά συγκεκριμένα προβλήματα. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Thank Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να είστε σύντομος κύριε Ντόσκης Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ πρόεδρε, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Φυσικά και θα τα λάβω αυτά υπόψη. Θα μελετήσω εις βάθος τα όσα είπανε για να τα εντάξω αυτά στην έκθεσή μου και σας διαβεβαιώ δε ότι θα προσπαθήσω σκληρά να μην αλλάξει η ουσία, η σπονδυλική στήλη της ε, έκθεσης, αλλά ταυτόχρονα να αφήσω περιθώριο για διαπραγματεύσεις, για συμβιβασμούς για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανησυχίες όλων των συναδέλφων. Η πορεία συνεχίζεται. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί έχουμε και την αξιοπιστία, έχουμε ό,τι χρειάζεται, έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Να, αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας, οπότε γι' αυτό και νομίζω ότι τελικά θα είναι δυναμική, θα είναι φιλόδοξη αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και εδώ κλείνει για αυτό το θέμα η συζήτηση και τώρα έχουμε την αναθεώρηση της στρατηγικής ΕΕ στον τομέα δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτή είναι η τελική συζήτηση για να καλύψουμε και τις τροπολογίες. Σκοπό αυτής της ε, έκθεσης είναι το πώς θα προτάξουν τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά και την πρόσφατη σφαιρική αναθεώρηση της στατικής της Ένωσης. Αυτό βεβαίως ε, ξεκινάει από την υπάτη εκπροσώπο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κυρία Άστον, και είπαμε ότι έχουμε ένα, μια στρατηγική πλαίσιο σφαιρικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Και έχουμε και το αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης. Ε, επομένως, θέλουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης να εφαρμοστεί ε, όπως πρέπει και αυτό να γίνει σε μια αρμονική συνεργασία με την εξωτερική υπηρεσία ε, και τα, τα, τα, μέλη, κράτη-μέλη, το, τον κύριο Λαμπρινίδη, το, τον ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα πριν δώσω εις, ε, τον εισηγητή το λόγο θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι 6 ενδεκάτου θα γίνει η ψηφοφορία. Κύριε Ταβάρης, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε το κείμενό σας. Thank you very much, Mr. President. Um, well, as, as you yourself as... Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, το σημείο κίνησης για την έκθεση αυτή είναι η κοινή δήλωση του ίδιου της είπα της εκπροσώπου και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού στις τρίτε χώρες εν ώψη της εφαρμογής του προγράμματος δράσης. Ξεκινήσαμε από μια πρώτη εξολόγηση για το πού βρισκόμαστε, την κατάσταση πρόοδου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι φτάσαμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα θα έλεγα ή μάλλον ένα πρώτο σημείο κίνησης που είναι το εξής. Η Ένωση βρίσκεται στα, σε μια φάση διπλής, ε, υποδιπλή ένταση. Δηλαδή, ταυτόχρονα ε, αποκτούμε περισσότερες αρμοδιότητες ε, και ταυτόχρονα από θεσμικής άποψης συγκεντρώνουμε νέες Αρμοδιότητε όσον αφορά το τομέα της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε την ύπατη εκπρόσωπο και τον ε, ε, ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε δηλαδή από μια πλευρά περισσότερες φιλοδοξίες και ευρύνουμε διευρύνουμε το φάσμα δράσης μας από θεσμικής άποψης, αλλά ταυτόχρονα όμως η πραγματικότητα είναι πιο δύσκολη. Ε, και γιατί γιατί υπάρχει η δημοσιονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συγκεκριμένα, αλλά και όσον αφορά την ε, αντίληψη περί Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν έχουμε το ίδιο βάρος, επιρροή, ε, κύρος ε, όπως παλιότερα. ξεκολουθούμε να έχουμε φυσικά επιρροή, αλλά η αίσθηση είναι διαφορετική. Και επίσης η ισορροπία δυνάμεων στον κόσμο φαίνεται να αλλάζει. Αν θέλετε λοιπόν υπάρχουν δύο πρόσφατα γεγονότα που νομίζω ότι επηρεάζουν αυτή την άποψη. Καπ' τη μια έχουμε την Αραβική Άνοιξη και το γεγονός ότι δεν, μπορούσαμε, δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε την Αραβική Άνοιξη και κατά κάποιο τρόπο προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε και να παίξουμε επικοδομητικό και χρήσιμο ρόλο. Ενώ ταυτόχρονα η ίδια η Ένωση, και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο, έχει αντιμετωπίσει αρκετές ε, συνέπειες της οικονομικής κρίσης και το βλέπουμε αυτό σε κάποια κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η ευάλωτος χαρακτήρα κάποιων ε, ε, κρατών λόγω της δημοσιονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα τα κατέστησε πιο, πιο, πιο ευάλωτα σε αγορές, εξαγορές από τρίτες χώρες, τρίτες χώρες όμως όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. We do not to, to, to... Τι πιστεύουμε εμείς. Εμείς δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε ε, όσον αφορά τις φιλοδοξίες. Πρέπει να ακολουθήσουμε ε, τις προτεραιότητές μας και τη θεσμοθέτησή τους αλλά ταυτόχρονα να τις ε, δεσμεύσουμε σε ένα μια εργαλειοθήκη που να είναι διακριτική, κατανοητή από την άλλη πλευρά η Ένωση πρέπει να δείξει κάποια ε, ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο ε, Ε, στον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργεί. Να ξέρουμε δηλαδή τι θέλουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, έξω κόσμος βέβαια. Ε, να δούμε λοιπόν το δεύτερο επίπεδο που είναι το επίπεδο της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Ένωση και τους θεσμούς της και το τρίτο επίπεδο είναι το δικό μας επίπεδο, το επίπεδο των διαθεσμικών σχέσεων μέσα στην Ένωση και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο ως ένα σώμα που έχουμε αναπτύξει με τα χρόνια ένα μεγάλο, μια μεγάλη παράδοση όσον αφορά τη δουλειά για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ελπίζουμε ότι θα ε, είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Έχουμε κάνει διάφορες προτάσεις. Μια από τις προτάσεις είναι ήδη υπό εξέλιξη, που είναι η δημιουργία ενός μια μιας ομαδα ομάδας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο και την Κομισιόν, ακριβώς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εργασία εδώ και κάποιου μήνε. με πολύ επικοδομητικό έργο. Αυτό που προτείνουμε είναι να τυποποιηθεί, να επισημοποιηθεί αυτή η ομάδα επαφής και να δουλεύουμε τακτικά σε αυτήν ώστε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Υπάρχουν επίσης κάποιες προτάσεις για συνέχεια γιατί έχουμε ένα μέγα πρόβλημα στο Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που δίνονται στα ίδια μας τα ψηφίσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις αντιπροσωπείς μας επιτόπου που μεταβαίνουν δηλαδή για να αξιολογήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες. Θα πρέπει να αναλάβει κάποιος να είναι υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε μόνιμη επιτροπή των, ανθρωπίνων, των, Ευρωκοινοβουλίου και αυτό να παρακολουθεί και τη συνέχεια που δίνεται στις επισκέψεις αυτές. Τρίτον, πρέπει με την νέα ε, εργασιακή σχέση που θα έχουμε τώρα με τον ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να δούμε και τη σχέση μας με τον εξωκόσμο. Δηλαδή έγινε μια πρόταση για μια συνέλευση νέων από τον αραβικό και τον ευρωπαϊκό κόσμο γιατί ένα από τα διδάγματα είναι ότι δεν ξέρουμε τις κοινωνίες, δεν τις γνωρίζουμε τις κοινωνίες που μας, που, με τις οποίες γειτονεύουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή ΑΦΕΤ που κάνει τη σημερινή συζήτηση. Έχουμε λάβει 147 τροπολογίες. Τις έχω μελετήσει όλες, σχεδόν όλες είναι ε, αποδεκτές, εμπίπτουν στο φάσμα των πιθανών ε, συμβιβαστικών τροπολογιών που πιστεύω θα είναι γύρω στις 20-25 με τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι σκιώδεις εισηγητές και άλλοι συνάδελφοι όπως και εσείς ο ίδιος. Ε, κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες δεν εμπίπτουν ε, στο πεδίο των συμβαστικών θα συστήσω να τις περιψηφίσουμε. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχει ευρεία συνένεση για την έκθεση αυτή. Θα γίνει μια συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε τις συμβιβαστικέ και είμαι ανοιχτός σε προτάσεις και σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Συμβολή των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Κίνγκα Γκάλ είναι η σκιώδης εισηγήτρια ε, του ΕΛΚ. Δεν είναι εδώ και μου ζήτησε ακόμα από μένα, και πάλι μάλλον από μένα, να παρουσιάσω τη δική της παρατήρηση. Συμμετείχε στις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής όπου εξετάστηκε το σχέδιο της έκθεσης σε αυτές τις ε, συνεδριάσεις παρουσίασε τα σχόλιά της ε, και τις παρατηρήσεις της σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης, ωστόσο λόγω του ότι έλαβε ε, τροπολογίες πλήρως μεταφρασμένες μόνο σήμερα, μάλλον προχτές την Δευτέρα και την Τρίτη έπρεπε να μεταβεί στο συνέδριο του ΕΛΚΕ στο Βουκουρέστι, δεν μπόρεσε να τις μελετήσει εις βάδος ακόμη. Ε, προσβλέπει στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών, των ε, σκιωδών, συγγνώμη, ώστε να εξετάσει τις τροπολογίες και να βρεθούν έτσι οι κατάλληλες συμβιβαστικές. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ζητήσω από τους υπόλοιπους ομιλητές να είναι σύντομοι και επί γιατί έχουμε ε, διακεκριμένο ε, σήμερα η κυρία Γκόμες. Εγώ μιλώ εξ ονόματος του Σκιώδου, ε, εισηγητή μα του κύριο Ρέιμον Ομπιόλ, που δεν μπορούσε να είναι παρόν. Θέλουμε να συγχαρούμε τον εισηγητή, τον κύριο Χούι Ταβάρες, για την εξαιρετική του εργασία. Ε, είναι πολύ καλό σημείο κίνησης για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις στον τομέα αυτό δουλέψαμε για τις τροπολογίες με στόχο να τονίσουμε κάποια θέματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά για μας Όπως είπε ο κύριος Ταβάρες, θα πρέπει να επιμείνουμε στα διδάγματα που αποκαμίσαμε από την Αραβική Άνοιξη, να αλλάξουμε τις προτεραιότητες και να θεσπίσουμε ένα πραγματικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. ΜΚΟ, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώσεις νεών, νέων και γυναικών που έπαιξαν φανταστικό ρόλο, αλλά επίσης πολιτικά κόμματα, συνδικάτα και ούτω καθεξής αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα απόλυτη για μας και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα από όσα έχουμε ήδη κάνει, κατά τη γνώμη μου. Έπειτα μέσα στο πλαίσιο των θεσμικών ε, οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών και συνεργασία μεταξύ τους μπορούμε να κινηθούμε. Ελπίζουμε λοιπόν πολλά από τον ε, ε, νεοδιοριστέντα ειδικό εκπρόσωπο κύριο Λαμπρινίδη που γνωρίζει τόσο καλά τις συνήθειές μας εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και το πώς λειτουργούν τα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσει πραγματικά να πετύχει πράγματα. Τρίτο, συνοχή ε, στις πολιτικές μας. Σε ολόκληρο τον κόσμο συνοχή των πολιτικών εκτός και εντός συνόρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί προσχάρουν τις ίδιε μας, τις αξιοπιστίες αλλά και τις αποδοτικότητάς μας. Και θα ήθελα να πω, ο κ. Ζωφή το τόνισε, ποιες ότι οι επιπτώσεις της ε, οικονομικής κρίσης είναι σημαντικές εγώ θα ήθελα αυτό να το μεταφράσουμε ως μια, μια ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της εταιρικής ε, κοινωνικής ευθύνης και ευθύνης των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για τα διδάγματα που πρέπει να αποκομίσουμε από αυτή την κρίση. Ξέρουμε και πολλοί από εμά πιέσαμε υπέρ της δημιουργίας του φόρου για τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ούτω καθεξής και αυτό θα είναι σημαντικό όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις τις οικονομικές αλλά αυτές θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις σχέσεις μας για με τις τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ειδικά αυτές τις χώρες που για τις χώρες που κυβερνώνται από διεφθαρμένες ελίτ που κρύβουν τα κέρδη τους στις δικές μας τράπεζες. Τέλος, δείκτες και ειδικά ορόσημα για τις ε, στρατηγικές σε χώρες όπου έχουμε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια η Κίνα κατέχει την πρώτη θέση. Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη επισημότητα σε αυτή τη ε, συζήτηση μέσω της συζήτησης που συνδέεται με τούτη τη στρατηγική, την αιτήσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Ευχαριστούμε κύριε Κοπά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική, ε, το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης, το οποίο βεβαίω αποδίδει τη σωστή σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία πρέπει να είναι στο κέντρο όλων των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχέσεων τη Ένωση με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων τομέων τη εξωτερική δράση τη Ένωση και να πιέσουμε για την εφαρμογή των ρητρών δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να μιλήσω για την έννοια της αμοιβαία λογοδοσία μεταξύ τρίτων χωρών Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών. Εμεί οι ίδιοι πρέπει να αποτελούμε παράδειγμα όταν μιλάμε για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Πρέπει να κοιτάξουμε και προ το εσωτερικό, στα του οίκου μα πριν ασκήσουμε κριτική στου άλλου το να υπάρχει επίσης συνοχή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών έχει κρίσιμη σημασία, γι' αυτό στηρίζω και τις αναφορές της σχετικές στο σχέδιο έκτασης. Με την ίδια λογική κατέθεσα και χαίρομαι που το έκαναν και άλλοι συνάδελφοι πολλέ τροπολογίες για να λάβουμε υπόψη την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές επιχειρήσεις αντικατοπτρίζουν το επίπεδο του πολιτισμού μας και έχουν επίσης ευθύνες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ, τα κράτη-μέλη της Ένωσης πρέπει να αναπτύξουν δικά τους εθνικά σχέδια για, για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αυτών αρχών και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε και οι χώρες εταίροι να τηρούν τα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο ο κ. Σταβάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τις ε, συναδέλφου, ε, τι κυρίες Κόμε και Κοπά και εσά που εκπροσώπησατε την κυρία Γκάλ. Δεν έχουμε χρόνο, βλέπω την κυρία Υπουργό και τον κύριο Πρέσβη. Θα επικεντρωθώ στο ζήτημα τη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι κρίσιμο. Καλωσορίζω τι ε, τροπολογίε που κατατέθηκαν στην έκθεση και νομίζω θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Είμαι υπέρ θεωρώ πως ε, το να να καταφέρουμε σωστά το ζήτημα των ε, επιχειρήσεων και των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σημαντικό και για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής γενικώ και για αυτά τα οποία θέλουμε να δούμε και στον κόσμο όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και τους άλλους τομείς που έχουμε προβλήματα πρωτογραφών που δεν εφαρμόζονται περιβαλλοντικών κτλ. Οπότε θεωρώ πως το γεγονός πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν ε, συμπεριφέρονται ε, σωστά και το ότι δεν, δεν επιβάλλουμε τη σωστή συμπεριφορά έχει σε εμάς, όχι μόνο στην αξιοπιστία μας, στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στην δική μας οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Αν δεν παίρνουμε λοιπόν σοβαρά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, νομίζω πως θα καταλήξουμε στην ίδια βραχυπρόθεσμη λογική που παριστάνει Ορισμένε φορές πως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απλά παρακολούθημα των λοιπόν πολιτικών αντί για κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και για ανθρωπιστικού, αλλά και ρεαλιστικούς λόγους. Συμφωνούμε νομίζω λοιπόν και αναμένω τις ε, συναντήσεις μας την ερχόμενη εβδομάδα για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ κύριε Ταβάρης. Περνάμε τώρα στην ενημέρωση από την κυρία Κοζάκου Μαρκουλή Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, εκ μέρους της ε, Κάθερινάς, Άστον Αντιπροέδρου της Επιτροπής και ΥΠΑ της εκπροσώπου, σχετικά με τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 15ης Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ και κύριε Βημό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι είχατε την καλοσύνη να περιμένετε και σας ευχαριστώ και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων της Επιτροπής για το ότι είστε στην διάθεση της Επιτροπής για να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών που έλεγε χώρα στην αρχή της εβδομάδας. Το Συμβούλιο συζήτησε αρκετά σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα την Συρία και την ε, δραματική κατάσταση στη χώρα αυτή η οποία δεν μας ανησυχεί απλώς αλλά πρέπει να μας κινητοποιήσει για να δράσουμε και να δράσουμε γρήγορα και απελεί βεβαίως και την ασφάλεια της ε, χώρας σας κατόπιν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γνωρίζουμε πώς οι διαπραγματεύσεις έχουν αποτύχει στο να δώσουν αυτά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο θέλει να διατηρήσει αυτή τη διτή προσέγγιση, να συνδυάσει δηλαδή τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με σκληρότερες κυρώσεις. Συζητήσατε και το Μαλί και την ανάγκη να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και η δαφική αικαιρεότητα αυτής της χώρας. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε λοιπόν τι προγραμματίζει να κάνει το Συμβούλιο και πώς σκοπεύει να στηρίξει τον ΟΗΕ υπό το φω τη πρόσφατης έντολη τη Ευρωπαϊκής Ένωση και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης η Λευκορωσία μας απασχόλησε μαζί με τις άλλες εξελίξεις της περιοχής. Δεν έχουμε λοιπόν πάρα πολύ χρόνο, οπότε σας δίνω αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής. Είναι ευχαρίστηση και τιμή να συναντώ σήμερα. Εξ ονόματος της είπα της εκπροσώπου και αντιπροέδρου της Επιτροπής της Βαρόνης ε, Άστον για να σας αναφέρω τα όσα έγιναν στο Συμβούλιο Εξωτερικών στις 15 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο ήταν ε, ένα επιτυχημένο και παραγωγικό συμβούλιο. Το βράδυ της 14ης το Συμβούλιο είχε δείπνο με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Συζητήσαμε διμερεί ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, το εμπόριο, ο συνεταιρισμός για τον εξυγχρονισμό σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών και θεωρήσεις διαβατηρίων και πάρα πολλά διεθνή ζητήματα όπως τη Συρία, το Ιράν και το Μαλί. Ήταν μια μακροσκελής και έντονη συζήτηση κατά την οποία κάθε πλευρά εξέθεσε τα επιχειρήματά της με ειλικρίνεια και σοβαρότητα. Συνολικά χάρη στην καλή ατμόσφαιρα που επικράτησε, η ορμή ε, της ε, κρίσιμης αυτής εταιρικής σχέσης ε, διατηρήθηκε και έτσι θα ε, προετοιμάσουμε καλύτερα τη Σύνοδο Κορυφής με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο. Το πρωί της Δευτέρας αποφασίσαμε όσον αφορά την ε, τελετή απονομής ε, του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάσουμε μια σύντομη δήλωση που βεβαίως δημοσιοποιήθηκε μετά το Συμβουλίο. Θεωρούν πως η αναγνώριση του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μία πρόσκληση για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για την ειρήνη και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών και να προσπαθήσουμε να γίνει η εξωτερική δράση πιο συνεκτική, συνολική και αποτελεσματική. Αυτό ήταν απευθεία από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Κατόπιν, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης μας απασχόλησε ήταν το μαλή. Η κατάσταση εκεί πέρα εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες σοβαρές το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε την περασμένη Παρασκευή ένα δεύτερο ψήφισμα το οποίο περιλαμβάνει πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει βοήθεια και εμπειροκνομοσύνη για να στηρίξει τις ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας του Μαλή. Για το σκοπό αυτό υιοθετήσαμε συμπεράσματα του Συμβουλίου που ζητάνε μια συνολική διαχείριση της κρίσης, μια στρατιωτική αποστολή ΚΕΠΑ για αναδιάρθρωση και επανεκπαίδευση του στρατού της χώρας αυτής. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε μια κοινή ανάλυση της απειλής που υπάρχει στην περιοχή, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο από την αστάθεια, την τρομοκρατία και το διεθνές έγκλημα οι στόχοι μας είναι σαφείς. Να επανέλθει το κράτος δικαίου και δημοκρατική κυβέρνηση η οποία θα ελέγχει όλη την επικράτεια της χώρας. Πρέπει να συνεργαστούμε επίσης στενά με τον ΟΗΕ, την Αφρικανική Ένωση και την ΕΚΟΒΑΣ, κάτι το οποίο τονίσαμε. Και ο ορισμός του Ρωμάνο Πρόντι ως ε, ειδικό πεσταλμένου του ΟΗΕ στο Σαχέλ ήταν κάτι το οποίο καλώς ορίσαμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε ε, στο ζήτημα αυτό στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Κατόπιν συζητήσαμε την κατάσταση στη Συρία. Η άμεση προτεραιότητα παραμένει βεβαίως το να σταματήσουν οι, ε, να σταματήσουν Κυρίως αυτό τονίσαμε. Επίσης, ε, υιοθετήσαμε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που στοχεύουν το καθεστώς και όχι τους πολίτες. Επίσης, τονίσαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανισχύει βαθύτατα από το πώς θα διαχυθεί η κρίση αυτή στις γειτονικές χώρες και καταδικάζει τον βομβαρδισμό της τουρκικής επικράτειας από τις συριακές δυνάμεις καλούμε τους πάντες να αποφύγουν την κλιμάκωση. Καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές και οι πολιτικές προσπάθειες, το Συμβούλιο εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις προσπάθειες του ΟΗΕ, του Αραβικού και του απεσταλμένου τους που είναι από με τον Αραβικό Σύνδεσμο του Λαχτάρ Μπραχίμι. Ταυτόχρονα ο χειμώνας ο οποίος έρχεται καθιστά όλο και πιο σημαντική την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κυρία Γεωργίευα μας ενημέρωσε για την σχετική βοήθεια. Ως ο μεγαλύτερος δωρητής με κονδύλια τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 230 εκατομμυρίων ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών σε αυτό το μέτωπο. Αλλά πρέπει να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερε προσπάθειε, ακόμα και σε γειτονικέ χώρε οι οποίε φιλοξενούν μεγάλο αριθμό Συρίων προσφύγων ή ε, ερχόμενοι σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών στην ίδια τη Συρία. Όσον αφορά την Αίγυπτο, η υπατή εκπρόσωπος μας ενημέρωσε για τις ε, προετοιμασίες της ε, συνεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου 12 Νοεμβρίου και βεβαίως ε, της ε, μονάδας δράσης για το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει να ενθαρρύνει τη διαδικασία μετάβασης και να φέρει σε επαφή πάρα πολλού ενδιαφερομένους. Επίσης απαντά στις κύριες δραστηριότητες της Αιγύπτου που αφορούν επένδυο, εμπόριο και ανάκαμψη του τουρισμού όπως βέβαια και σε προηγούμενες μονάδες δράσης, η εκπρόσωπος ε, προσκάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση. Επίσης, συζητήσαμε την διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Εδώ πέρα είμαστε ενωμένοι στον στόχο του να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων με στόχο να υπάρξει μία λύση. Δύο κρατών μετά από διαπραγματεύσεις η οποία θα προσφέρει ειρήνη και σταθερότητα και για τις δύο πλευρές. Για το Ιράν συμφωνήσαμε σε νέα περιοριστικά μέτρα που εστιάζονται σε τέσσερις κυρίως τομείς. Χρηματοοικονομικά, εμπόριο, ενέργεια και μεταφορές. Τα μέτρα αυτά είναι σχεδιασμένα για να στοχεύσουν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και στα έσοδα του καθεστώτος που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα αυτό δεν έχουν στόχο τον Ιρανικό λαό. Η απόφαση αυτή στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιράν για να απαντήσει στις σοβαρές ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την φύση του πυρηνικού του προγράμματος και να απαντήσει στην πίεση για ε, επικοδομητικές επαφές. Ταυτόχρονα το Συμβουλίο επαναβεβαίωσε στα συμπεράσματα τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εργαστούμε για μια διπλωματική λύση στο ζήτημα του Ιράν μέσω μιας δικασίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα βασίζεται στις αρχές μιας σταδιακής προσέγγισης και της αμοιβαιότητας. Οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Επαφίεται στο καθεστώς του Ιράν να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα επιτρέψουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης όσον αφορά την αποκλειστικά ειρηνική φύση του πυρηνικού τους προγράμματος. Οι τρεις συν θα συνεχίσουν να πιέζουν το Ιράν για να έρθει σε διάλογο ως με βάση αυτή την διτή προσέγγιση. Στο μεσημεριανό συζητήσαμε την ανατολική γειτονία, εστιαζόμενοι κυρίως στην πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία και τη Γεωργία μετά τις εκλογέ. Για τη Λευκορωσία συμφωνήσαμε με την ανάλυση πως δεν υπάρχει πραγματική αλλαγή. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε ενωμένοι στην πολιτική μας για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους. Θα επιμείνουμε λοιπόν στην πολιτική μας της κριτικής εμπλοκής, θα ασκούμε κριτική στην έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα εμπλακούμε με την κοινωνία των πολιτών και την πολιτική αντιπολίτευση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και η παράταση των περιοριστικών μέτρων τονίζουν αυτή την προσέγγιση. Όσον αφορά τη γεωργία, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην μετεκλογική φάση. Πρέπει να διασφαλίσουμε συνέχεια στο, στα θέματα τα οποία μας απασχολούν με τη γεωργία και είναι αρκετά και να παραμείνουμε σε επιφυλακή καθώς η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήσαμε τονίζουν αυτό το γεγονός. Η υπατή εκπρόσωπος ανακοίνωσε πως είχε ζητήσει από τον Επίτροπο Φίλε μαζί με την ε, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Κέλκε Σμιτ να επισκεφθούν τη Γεωργία, να συναντηθούν με τις δύο πλευρές και να ενημερώσουν την νέα κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη συνεργασία με τη Γεωργία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πραγματοποιούνται αυτές οι επισκέψεις. Ο Επίτροπος Φίλε και η κυρία Σμιτ ε, νομίζω χτες το βράδυ αναχώρησαν και λαμβάνει η χώρα σήμερα η συνάντηση αναμένουμε την συζήτηση που θα ε, έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τη Λευκορωσία και για τη Γεωργία. Αυτά είχα να σας πω. Όπως είπα και στην αρχή, υιοθετήσαμε συμπεράσματα ε, για την Συρία, το Ιράν, την Λευκορωσία, τη Γεωργία και η το Που βεβαίω είναι στη διάθεσή σας. Είμαι και εγώ στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Για αυτήν την ολοκληρωμένη σας ε, παρουσίαση όσον αφορά τους προβληματισμούς αλλά και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνάδελφοι, τώρα μπορείτε να αποβάλλετε τις ερωτήσεις σας ή τις παρατηρήσεις σας. Παρακαλώ προσπαθήστε να είσαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται, ούτως ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν. Και να έχει χρόνο και κύριε Υπουργός να μπορέσει να απαντήσει στη συνέχεια. Κύριε Ντεκάτσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία. Τρεις ερωτησούλες. Πρώτα πρώτα μας αναφέρει τον κύριο Λαυρόφ και την συνάντηση κορυφής ΕΕ Ρωσίας υπήρξε στροφή της Συρίας ή τέλο πάντων υπήρξε στροφή της Ρωσίας όσον αφορά το Συριακό. Για πετε μας γιατί στα συμπεράσματα δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Δεύτερη ερώτηση. Μας είπατε με δύο λόγια το τι γίνεται με το Παλαιστινιακό, με, με το Μέσα Ανατολικό. Τι έγινε με τον ε, Αμπά τον τι έγινε με το ψήφισμα. Ε, είναι κάπως διφορούμενα ε, τα όσα διατυπώνονται στο ψήφισμα τώρα για το Ιράν. Βεβαίω. Για τον εμπλουτισμό σε ουράνιο βρίσκουν πολλές δικαιολογίες οι Ιρανοί. Καλά εντάξει υπάρχουν και οι ιατρική σκοπή του εμπλουτισμού, αλλά έχουν ξεπεράσει τα προηγούμενα όρια, γιατί μου τα εξήγησε και με ο πρέσβης, για τα ραδιοϊσότοπα, ότι γίνονται προσπάθειες Γίνονται διαβήματα πρώτα τα προς Ρωσία, μετά προς Βραζιλία. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αλλά η Ευρώπη πώς βλέπει το θέμα. Τι λέτε για το Ιρανικό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκόμες. Merci, Madame le Ministre. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω, να σας ρωτήσω κάτι για την αποστολή στο Μαλί. Την αποστολή της ΚΕΠΑ. Για πέστε μας. Θα θέλετε τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν την αποστολή. Παρά την οικονομική κρίση. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε πόσο ατυχής ήταν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια γειτονική χώρα όπου και εκεί υποτίθεται ότι θα αντιμετωπιζόντουσαν τα προβλήματα τα οποία τώρα θέλουμε να επιλύσουμε στο Μαλί. Μίλω για την Γουινέα Μπισά. Και εκεί θέλαμε να υπάρχει αναδιάρθρωση του στρατού, όμως να πρετανεύσει το κράτος δικαίου, να καταπολεμηθούν τα ναρκωτικά, οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Χειροτέρεψαν τα πράγματα. Τίποτα δεν έκανε η Ένωση. Φοβάμαστε επομένω ότι θα γίνουν τα ίδια και με το Μαλί. Και βάσει τόσο δεν πρέπει να φλούμες, σχέση με το τι ισχύει τώρα στη Γουινέα Μπισάου. Τι θα γίνει, θα ζητούν αυτά στο Συμβούλιο. Σας ρώτησε η Βερονίκ για τη Συρία, αλλά έχω εγώ και μια άλλη ερώτηση σχετικά. Έρχεται ο χειμώνας και έγινε κάποια σοβαρή συζήτηση για το πώς μπορούμε να έχουμε κάποιο είδους ε, ασφαλείς περιοχές για ανθρωπιστικούς λόγους, όχι εδώ στη Συρία, αλλά στη γειτονική Τουρκία ή αλλού και εξασφάλισε φυσικά αυτών των φυλάκων, των ανθρωπιστικών. Και για το Μεσανατολικό, η Βερονίκη επίσης ρώτησε τι γίνεται με την Παλαιστίνη στο ΟΗΕ. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε Τι είναι στο Συμβούλιο όσον αφορά την ενευτική διαδικασία. Προχωράει. Δεν είναι εντύπωση στο Συμβούλιο ότι είναι υπέρ της Συμφωνίας ΣΑΚΑ που δεν συνάδει προς τους σκοπούς τους ενευτικούς. Σας ρωτώ γιατί εκτός από το Συμβούλιο αυτό έχει σημασία για τη χώρα σας και για την Τουρκία. Μια που πρόσφατα ο κύριος Μπαρόσο όρισε έναν εκπρόσωπο για να ασχοληθεί με το Κυπριακό. Τι λέτε γι' αυτά. Κύριε Χουντή. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Υπουργό για την ε, συμμετοχή της στη σημερινή μας συνεδρίαση για την ανάλυση που έκανε στα συμπεράσματα της Συνόδου. Σπέβδω να πω ότι ερωτήσεις αλλά και παρατηρήσεις σχετικά με αυτά που είπε και με αυτά που έχω πληροφορηθεί δεν την αφορούν προσωπικά, έχουν μια γενικότερη σημασία γιατί καταλαβαίνω ότι απηχεί μας έδωσε τα συμπεράσματα ε, της κυρίας Άστον ή του Συμβουλίου γενικώ. Επομένως οι παρατηρήσεις που θα πω και ερωτήσεις δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα για την Υπουργό. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Είναι πολύ γενική και σε σχέση με τα θέματα της, ε, των εξεγέρσεων στις αραβικές χώρες, τη Συρία σήμερα και το πρόβλημα του Ιράν, τα δύο τελευταία από ό,τι κατάλαβα συζητήθηκαν. Πείτε μου σας παρακαλώ μια γενική εκτίμηση αν μπορείτε. Η Ευρώπη κάνει ό,τι, είναι δυνατόν να λυθούν με ειρηνικό τρόπο αυτά τα θέματα. Σπέβδω να πω ότι πιστεύω πως δεν το κάνει. Και επιτρέψτε μου και μια παρατήρηση ίσως επίκαιρη. Πέρα από την ουσία, στο συμβολικό η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το φιλιρινικό ρόλο αναμετριέται με την αμφιλεγόμενη για πολλούς απόφαση απονομής της του βραβείου Νόμπελ. Ε, θα αναμετριέται, αν ήταν πιστική, αν έκανε πράγματι. Θα έλεγα εγώ έτσι, αν πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερνε να αντιμετωπιστούν με δίκαιο τρόπο χρονίζοντα προβλήματα που την αφορούν πολύ άμεσα όπως, θα, όπως είναι το, το Παλαιστινιακό και το Κυπριακό τότε αν γινόταν ξανά ψηφοφορία ναι βραβείο Νόμπελ. Αλλά τώρα είναι συζητήσιμο. Συρία λοιπόν και Ιράν. Και έρχομαι πιο συγκεκριμένα για να γίνω πιο κατανοητός. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει καλή ανάλυση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της εξέγερσης στις αραβικές χώρες ή αν θέλετε και της σημερινής κατάστασης στη Συρία. Το ερώτημα που θέλω να θέσω ε, πρέπει να λυθούν ειρηνικά χωρίς παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ιδιαίτερα το Συριακό. Πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο των Υπουργών, την ανάμιξη της Τουρκίας και την προσπάθεια να αποκτήσει πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Η ανάμειξη της Τουρκίας από τη μια, ο έτσι και αλλιώς παρεμβατικός ρόλος του, του Ισραήλ σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Δεν δημιουργεί, κυρία Υπουργέ, νέες αντιφάσεις σε αυτή την κατάσταση και κινδυνεύει η ανάφλεξη να πάρει γενικότερες συνέπειες και η διάχυση να κινδυνεύσει σε όλη την περιοχή. Νομίζω καταλαβαίνετε ορισμένε πλευρέ, δύο πλευρέ θα πω και δεν θα σα κουράσω. Ε, μέτρα και αντίπεινα σε βάρο του Ιράν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικέ χώρε ε, ενεργειακή επάρκεια σε πολλέ χώρε, στη χώρα μου το δημιουργεί. Επομένω, ε, πρέπει να τη αυτή τη συνέπεια. Στρατιωτική επέμβαση στη Συρία θα δημιουργήσει νέα κύμα, νέο κύμα συγγνώμη, προσφύγων που θα πάνε προς την Ευρώπη, θα περάσουν από την Ελλάδα, μιλώ και από αυτή την ελληνική πτήση. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Επομένως, ε, ε, θέλω να πιστεύω ότι τα συζητάτε ή πείτε μου ότι σας ανησυχούν ή ότι, εν πάση περιπτώσει για να μην σας κουράζω περισσότερο, ότι τέτοιες πλευρές στην ανάλυση των, αυτής της κατάστασης ε, σίγουρα εξετάζονται και, εν πάση περιπτώσει, θα περιμένω λέω μια άποψη, την άποψη της ομάδας, πιο ενεργητική φιλιρινική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Mr. Sofokleus is the next speaker. Please. Ευχαριστούμε κύριο Σοφοκλέους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να καλωσορίσω την κυρία Υπουργό να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την σύντομη δήλωση όπως έχει κατατεθεί από το Συμβούλιο, δηλαδή η πρόθεση της ειρήνης και η εξωτερική δράση πρέπει να είναι πιο συνεχτική. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτή την γενική δήλωση. Επίσης πρέπει να πούμε ότι πολύ σωστά γίνεται μια αναφορά, μια περιγραφή σε ανοιχτά ζητήματα όπως είναι το Μαλή, η Συρία, η Αίγυπτος, του Παλαιστινιακών, Ιράν, Λευκορωσία και Γεωργία. Και επίσης η τοποθέτηση η οποία έχει κατατεθεί είναι στα πλαίσια της διεθνής έννομης τάξης του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού και Κεκτημένου και επίσης δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει για το ενδιαφέρον. Θα περιοριστώ όμως σε τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, αφορά την, την Συρία. Και ακούσαμε την κυρία Νάστον και στην Ολομέλεια, όπου έκανε μια περιγραφή, μια στήριξη κυρίως οικονομική και ανθρωπιστική προς την Συρία. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχει ένα, θα τολμήσω να πω, σχέδιο Β για τη Συρία, αφού καθημερινά με τις παρεμβάσεις σας και την παρουσία σας ε, δεν μειώνονται οι δολοφονίες. Καθημερινά έχουμε δολοφονίες. Αυξάνονται οι δολοφονίες. Αυξάνονται οι απειλές αυξάνεται η πιθανότητα μια σύραξη. Βλέπουμε την Τουρκία όπου επικίνδυνα, αν θέλετε, τοποθετείται και επίση Ρωσία, Κίνα, με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε τοποθετούνται. Υπάρχει ένα σχέδιο Β, δηλαδή πρακτικό, συγκεκριμένο το πώ θα υπάρξει ειρήνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Και το, το δεύτερο μου ερώτημα είναι το Παλαιστινιακό, δηλαδή το να τοποθετούμαστε περίπου ως ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση, ε, νομίζω το λέμε για πάρα πολλές δεκαετίες, ε, δύο κράτη, έννομη τάξη, διεθνές δίκαιο. Επίσης εδώ μπορούμε να σπρώξουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση με ένα πρακτικό συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει ένα σχέδιο. Και το τρίτο έγινε μια αναφορά από την συνάδελφο την κυρία Γκόμες για τον διορισμό εγώ λέω ενό τεχνοκράτη, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση, μεσολαβητή για να βοηθήσει στην προοπτική διαλόγου και λύση του κυπριακού προβλήματο. Η ερώτησή μου είναι με αυτή την ευκαιρία μελετάτε ή μπορεί να μελετηθεί να υπάρξει μια πολιτική προσωπικότητα χωρίς να μειώνω αυτή την προσωπικότητα, την τεχνοκρατική που μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες για να βοηθήσει. Αυτά είναι τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Σας γνωρίζω χρόνια κυρία Υπουργέ και ξέρω ότι δεν αποφεύγετε να απαντήσετε με έναν ευθύ και κυρίως ε, καθαρό τρόπο και πρακτικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Leinen. And then I'll give the floor to the Minister. Ευχαριστώ κύριος Λάινεν και μετά κύριε κυρία <laughs> Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε τη Γεωργία και είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται ενεργά με τις εξελίξεις σε αυτή τη χώρα. Η Γεωργία έχει μια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση που προετοιμάζεται και καλό θα ήταν να συναυθεί η συμφωνία, θα βοηθούσε τη χώρα. Το ερώτημα είναι πώς αξιολογεί το Συμβούλιο την νέα Προεδρία της Γεωργίας σε σχέση με τη Ρωσία. Και πέρα θα μπορούσαμε να έχουμε θετικές εξελίξεις καθώς η νέα κυβέρνηση ε, έχει μια καλύτερη συνεννόηση με τη Ρωσία. Να αναφερθώ και στα της Μέσης Ανατολής μιλήσατε για μια λύση δύο κρατών αλλά δεν, μπορούμε να, δεν κάνουμε τίποτα για τον ε, επικισμούς του Ισραήλ στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Δεν θα υπάρχει τίποτα για να υπάρχουν δύο κράτη σε λίγα χρόνια. Θα έχουμε ένα μόνο κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί αβοήθητη την ε, κατάσταση και δεν κάνει και αρκετά για να σταματήσει την ε, οικοδόμηση επικισμών, ίσως και με, μέτρα που θα δείξουν στο Ισραήλ πως δεν συμφωνούμε. Συρία και ο κίνδυνος μετάδοσης ε, στις γειτονικές χώρες, ε, κυρίως στην Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω τι κάνουμε για να εμποδίσουμε έναν πόλεμο εκεί πέρα Ε, γιατί από αψιμαχίες ε, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Λάινεν. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην ε, κυρία Υπουργό για να απαντήσει. Σα σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, υπήρξαν πολλές ερωτήσεις κάποιες νομίζω ταυτίστηκαν. Θα προσπαθήσω λοιπόν όσο μπορώ να απαντήσω με τρόπο συνολικό. Όσον αφορά την συνάντηση με τον κύριο Λαυρόφ, όπως είπα, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και για διμερή και για διεθνή ζητήματα και κυρίως τη Συρία, το Ιράν και το Μαλί. Για τη Συρία βεβαίως συμφωνήσαμε πως διαφωνούμε σε κάποια ζητήματα με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αυτό είναι γνωστό, αλλά θα πω πως έγινε μια καλή συζήτηση και ειλικρινής κατά τη διάρκεια του δείπνου. Και αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι πως ο κύριος Λαυρόφε επανέλαβε την, ε, τις θέσεις της ε, χώρας όσον αφορά το ανακοινωθέν της Γενέβης, ε, το οποίο είπε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης και δεν μπορώ να πω πως υπήρξε κάποια κίνηση προς την κατεύθυνση της σύγκλησης όσον αφορά τις διαφορές που έχουμε για τη Συρία αλλά και πάλι θέλω να επαναλάβω πως η συζήτηση ήταν επικοδομητική, ειλικρινής και όπως είπε και η ύπατη εκπρόσωπος ήταν μια καλή προετοιμασία για την Σύνοδο Κορυφής με τη Ρωσία για τη Μέση Ανατολή. Συζητήσαμε βεβαίως όλα τα ζητήματα το Συμβούλιο τον Μάιο υιοθέτησε ε, κάποια από τα πιο ε, έντονα θα έλεγα συμπεράσματα που έχει οδητήσει ποτέ έντονες θέσεις ε, για τους οικισμούς και την λύση των δύο κρατών που θέλουμε υπήρχε συζήτηση για την δήλωση του Προέδρου Αμπάς για ένα ψήφισμα που θα υποβληθεί αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γενική Συνέλευση αλλά θα έλεγα πως η συζήτηση κυρίως επικεντρώθηκε στο πως μπορούμε να είμαστε πιο επικοδομητικοί στο να ξανά ξεκινήσει η διαδικασία αυτό είναι το βασικό αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιο είναι το περιεχόμενο του ψηφίσματος που θα κατατεθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή. Οπότε ο στόχο είναι να ξαναξεκινήσει η διαδικασία και αυτό ήταν βεβαίως το αντικείμενο της συζήτησής μας. Για τους οικισμούς βεβαίως τους επικισμούς. Ε, νομίζω πως η θέση μας είναι σαφής και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στις δηλώσεις της ΥΠΑ Προσώπου εκπροσώπου. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς πως είναι απαράδεκτο και είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η θέση μας είναι σαφής και αν διαβάσει κανείς τα συμπεράσματα του Μαΐου η θέση αυτή επαναλαμβάνεται με τους ε, στεναρότερους όρους για το Ιράν. Και πάλι η θέση μας είναι σαφής και αντικατοπτρίζεται στα πρόσφατα συμπεράσματα. της Δευτέρας. Βεβαίω οι κυρώσεις δεν είναι πολιτική από ε, μόνες τους, δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι μέρος της δυτής αυτής προσέγγισης, όπως ανέφερα, με μια πολύ σημαντική διπλωματική πτυχή. Γνωρίζετε, πως είπατε, εκπρόσωπο έχει συναντήσεις με την Ιρανική πλευρά στην ε, διαδικασία 3 συν και ταυτόχρονα προσπαθούμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη και γίνονται σχετικές προτάσεις. Οπότε, η θέση του Συμβουλίου είναι σαφής, καταδικάζει την συνεχιζόμενη παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου και την επέκταση της δυνατότητας εμπλουτισμού και τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες βαρέως ύδατος. Σύμφωνα με το ψήφισμα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή λοιπόν είναι η θέση του Συμβουλίου. Όσον αφορά τώρα την αποστολή στο Μαλί, Βεβαίω. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπατε πρόσωπος είναι στη διαδικασία σύστασης ε, της αποστολής της ΚΕΠΑ. Είναι πολύ νωρίς να πούμε λοιπόν ποια θα είναι η απάντηση των κρατών Αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις σοβαρές ανησυχίες που εκφράστηκαν στα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου, εγώ θα έλεγα πως παρά την κρίση, παρά την οικονομική κατάσταση, η απάντηση από πλευράς κρατών μελών θα υπάρξει προσεχώς. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις ερχόμενες εβδομάδες η κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου, κυρία Γκόμες, είναι ιδιαίτερο ανησυχητική. Είχαμε χτες την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακροτηρίου, να συζητήσουμε την κατάσταση στη Γουινέα Μπισάου. Βεβαίως, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα το πράσινο ακροτήριο ε, λόγω της γειτονίας με τη χώρα. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες που γίνονται στη χώρα. Βεβαίως ο πληθυσμός υποφέρει από όλες αυτές τις εξελίξεις. Και αυτή είναι μια κατάσταση στην οποία το Συμβούλιο έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί στο παρελθόν και βεβαίως εξακολουθεί να μας ανησυχεί. Αλλά η κατάσταση στο Μαλή και η ευρύτερη κατάσταση στο Σαχέλ ανησυχεί ιδιαίτερα το Συμβούλιο Γι' αυτό και ελήφθη αυτή η απόφαση κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όσον αφορά το τα ανθρωπιστικά ασφαλή μέρη για τους, για τους ε, Σύριους πρόσφυγες ε, έγινε αυτή η πρόταση για τη δημιουργία τέτοιων ε, θυλάκων εντός της Συρίας μέσα στην ίδια τη χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν κοινή θέση για αυτή την πρόταση ιδιαίτερα γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, διότι είναι, κάτι, είναι, είναι άλλο να φτιάξει κανείς διαδρόμους ή ασφαλείς περιοχές σε... και άλλο είναι να μπορέσει να προστατεύσει όντως τον πληθυσμό που θα ε, πορευθεί προς τα εκεί. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ομοφωνία αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την ώρα. Φυσικά η ανθρωπιστική κατάσταση είναι εξαιρετικά ε, σοβαρή σκοτώνεται κόσμος καθημερινά. το σύνολο ξεπερνά τις 40.000, το σύνολο των θυμάτων. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να πάψει η βία και, και οι, τα ανθρώπινα θύματα. Το Συμβούλιο δίνει πλήρη στήριξη στην αποστολή του κυρίου Μπραχήμη, ο οποίος όπως ξέρετε τώρα κάνει διάφορες επισκέψεις στις χώρες κλειδιά, ξεκινώντας βέβαια με την ίδια τη Συρία, αλλά και με όλες τις γειτονικές χώρες η ύπατος εκπρόσωπος αλλά και πολλά κράτη-μέλη συναντήθηκα με τον κύριο Μπραχήμι στη Νέα Υόρκη στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης και φυσικά έχει την πλήρη μας στήριξη. Για την ΆΚΑ, τη συμφωνία ΆΚΑ, δεν υπάρχει κοινή θέση όπως ξέρετε στο Συμβούλιο. αλλά κάποια μεμονωμένα μέλη έχουν λάβει στεναρή θέση υπέρ της εφαρμογής των αποφάσεων για προϊόντα που προέρχονται από τα κατεχόμενα και από τους επικισμούς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινή θέση στο Συμβούλιο. Έγιναν δύο ερωτήσεις σε σχέση με την Κύπρο, το Κυπριακό και τον ορισμό ενός νέου εκπροσώπου του κυρίου Μπαρόζο. Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω αυτή την ερώτηση προσωπικά, γιατί βρίσκομαι εδώ υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου της ΣΥΠΑ της εκπροσώπου και ελπίζω ότι θα το κατανοήσετε αυτό. Δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω να απαντήσω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο ειλικρινής είμαι, αλλά νομίζω πως αυτή τη φάση δεν είναι η κατάλληλος χώρος. Μιλάμε για τα απορίσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και ευχαριστώ να συζητήσω μακρόν το Κυπριακό σε κάποια άλλη στιγμή ή διμερός με τους συναδέλφους. Τώρα, υπήρχε άλλο ένα ερώτημα το οποίο αφορά τις αραβικές χώρες, την αραβική άνοιξη και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πώς να το πω, ε, κάποιες ε, επικρίσεις, τέλος πάντων αμφιβολίες για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση άξιζε το Νόμπελ το οποίο της απονεμήθηκε. Σας επαναλαμβάνω. Προβήγαμε την Δευτέρα ως Συμβούλιο σε κάποια ανακοίνωση, ως Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ακριβώς για την απονομή του βραβείου Νόμπελ. Απονεμήθηκε λόγω των όσων έχει πετύχει σε όλη τη διαδρομή Ευρωπαϊκή Ένωση και για μας δεν στέκει καμία αμφιβολία για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα όραμα ειρήνης. Από τότε, από τότε που ξεκίνησε τη διαδρομή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαμε κανέναν πόλεμο. Αλλά έχουμε συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και στην ειρήνευση και εκτός των σύνορων της, της Ένωσης, της Ευρώπης. Φυσικά και αποτελεί μια ενθάρρυνση η απονομία αυτού του βραβείου, ώστε να συνεχίσουμε. Και οι ευθύνε μας είναι τεράστιες, όπως αναφέρατε. Έχουμε το Παλαιστινιακό, την Αραβική Άνοιξη και τι άλλε κρίσεις που σοβούν παγκοσμίω. βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μόνος παίκτη στην παγκόσμια σκακέρα. Και έχουμε περιφερειακές ε, ενώσεις κρατών, άλλες δυνάμεις. Προσπαθούμε εμείς να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο. Και πάντοτε σε συνεργασία με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς και με περιφερειακούς οργανισμούς. Και ακριβώς γι' αυτό και για τη Συρία είναι πάρα πολύ στενή συνεργασία με τον Αραβικό Σύνδεσμο θα έχουμε συνάντηση επομένω σε και συνδέσμο σε υπουργικό επίπεδο. Θα πρόκειται για την δεύτερη μόλις συνάντηση που έχει γίνει ποτέ. Θα γίνει στο Κάιρο στις 13 Ενδεκάτου. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία ούτω ώστε και τα δύο μέρη να κάτσουν και να συζητήσουν όλα όσα γίνονται νοτίως της Ευρώπης πολλά θέματα. Έχουμε αυτή τη, τη συνεχή αλλαγή, το συνεχή μετασχηματισμό αυτών των, των χωρών νότιου της Ευρώπης. Εμείς δεν θα πάψουμε τις προσπαθίες μας να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές <coughs> και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περαιτέρω και σε συνεργασία βεβαίω με τους άλλους οργανισμούς. Τώρα όσον αφορά το ρόλο της Τουρκίας Βεβαίω πρόκειται για μια χώρα που έχει δραματίσει και θέλει να συνεχίσει να δραματίζει ρόλο στην περιοχή. Αλλά δεν είναι η μόνη. Είναι σημαντική στην περιοχή. Βεβαίω υπάρχουν και άλλες σημαντικές χώρες στον αραβικό κόσμο που έχουν το ρόλο τους. Σας είπα και ο αραβικός σύνδεσμος θα πρέπει να του δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά τα ζητήματα, τα σχετικά με την Αραβική Άνοιξη, με τις ε, εξελίξεις που απορρέουν τέλος πάντων. I think I have, uh, I have covered. Νομίζω ότι εκάλυψα τις ερωτήσεις εκτός αν κάνω λάθος, οπότε μπορείτε να μου πείτε. Πάνω κάτω σας τα είπα όλα. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε για την επίσκεψή σας, για, για, για αυτήν την ειλικρινή συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε άλλα δύο θέματα στις μέσες διατάξεως ευχαριστώ που δεν έχετε κάτι να πείτε για τα διάφορα, οπότε σα ενημερώνω ότι η επόμενη συνάντησή μα πρόκειται να είναι έκτακτη συνεδρίαση τη Επιτροπή των Υποθέσεων την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη στο Στρασβούργο. Την Πέμπτη στο Στρασβούργο και όπου θα γίνει και η ψήφιση. Η ψηφοφορία από τι 10 μέχρι τι 11.30, την Πέμπτη την επόμενη εβδομάδα. Εξαντλήσαμε τη μέση διάταξη. Πέρα συνεδριάζω, σα ευχαριστώ.